Η κυρία Γιάννησεν από τους Φιλελευθέρους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για το νέο σας αξίωμα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο που επιτέλους έχουμε έναν πρόεδρο που αρχίζει την ώρα του. Ε, κοιτάξτε, η θέση μας ευθυγραμμίζεται με αυτή των άλλων δύο πολιτικών ομάδων και του κυρίου Κόλιτσεκ. Για τα διευρωπαϊκά δίκτυα θέλαμε να μιλήσουμε και για ιδιαίτερα πώς ε, προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα 500 επιπλέον εκατομμύρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας. Η είναι τα προγράμματα, αλλά δεν έχουμε επαρκή χρηματοδότηση. Οπότε η γραμμή μας κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να είναι να αποκαταστήσουμε όλα αυτά τα χρήματα που ε, έχει αποκτήσει επιπροσθέτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από εκείνο το σχέδιο ανάκαμψης για την ε, υπηρεσία ασφαλείας ε, της πολιτικής αεροπορίας. Θέλουμε να διευρυθούν τα καθήκοντα της υπηρεσίας και να χορηγήσουμε και τα πετούμενα κονδύλια γι' αυτό. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να έχει επαρκή χρηματοδότηση η υπηρεσία. Οι φιλελεύθεροι θεωρούν ότι υποστηρικτικέ δραστηριότητε για, για, για την πολιτική μεταφορών και για τα δικαιώματα των επιβατών έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και θέλουμε να αποκαταστήσουμε το προσχέδιο προϋπολογισμού, δηλαδή να καλύπτονται αυτές οι απαιτήσει μας. Πιλωτικά προγράμματα δεν προβλέπονται προς το παρόν. Έχουμε επιτύχει στις διαπραγματεύσεις επίσημα στην Επιτροπή Μεταφορών πάντως. Θα πρέπει να υποβάλουμε τροπολογίες πριν τις διακοπές. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να μεταφραστούν για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε για τις τροπολογίες το Σεπτέμβριο. Ε, ε, μάλλον δεν θα καταφέρουμε και πολλά πράγματα αυτή τη φορά. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι πράσινοι θέλουν ε, να κάνουν περισσότερα πράγματα για κάποια προγράμματα. και θα τους ε, στηρίξουμε γιατί έχουμε ήδη συνεργαστεί μαζί τους για κάποια θέματα. Μάλιστα κυρία Γένσεν, κανονικά πρέπει να έχετε ένα φάκελο από τη Γραμματεία για την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού και πρέπει να έχετε πάρει κανονικά και ένα φάκελο από την Επιτροπή για όλα τα προγράμματα που τρέχουν και πάνω πάνω είναι το τρένο του Σιδρού παραπετάσματος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ βέβαια δεν είμαι σε θέση να το σχολιάσω όπως καταλαβαίνετε και πάω στον κύριο Μάικλ Κρέμε, το συντονιστή των Πρασίνων. Μετά από τόσες φιλοφρονήσεις τι να πω, εγώ δεν έχω τίποτα να αντιτάξω. Βέβαια, το είπατε και χαίρομαι που μας υποστηρίζουν και οι φιλελεύθεροι και εσείς ε, το ε, πρόγραμμα αυτό. Στην έκθεση Λίχτεμπεργκερ με μεγάλη πλειοψηφία αποφασίσαμε στην Ολομέλεια για τα δύο δίκτυα να μην έχουμε μόνο το σιδηρόδρομο και ε, τους δρόμους και τα ε, αεροδρόμια αλλά και ε, τους διαφόρους ε, δρόμους ποδηλάτου και θα πρέπει και οικονομική υποστήριξη να υπάρχει. Ελπίζω να συμφωνήσετε γιατί καλές είναι διακηρύξεις αλλά θα πρέπει να βάλουμε και το χέρι στην τσέπη διότι αλλιώς δεν γίνεται. Τώρα, για τα οικονομικά προκύπτει τελικά ότι αυτά που φοβόμαστε επιβεβαιώνονται όταν αποφασίσαμε τον προπολογισμό. Τα βρίσκουμε μπροστά μας. Γιατί ποια ήταν η συνέπεια. Ακριβώς επειδή τα τελευταία χρόνια και δεκαετίες το Ταμείο ήταν μείον για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ήθελαν να αυξήσουν κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ ε, από το 2007-2013 το προϋπολογισμό και είπαμε τα διασυνοριακά ε, προγράμματα μέχρι 50% χρηματοδότηση. Για μας ήταν απολύτως σημαντικό γιατί για τα κράτη-μέλη τα μεμονωμένα οι παραμεθόριες ε, διαδρομές είναι λιγότερο ε, αποτελεσματικές και έχουν χαμηλότερο εθνικό ενδιαφέρον, αλλά έχουν για μας ενδιαφέρον ευρωπαϊκό. Γι' αυτό είπαμε μέχρι 20 δις και 50% χρηματοδότηση. Και είχαμε βάλει και προτεραιότητες των προτεραιοτήτων, όλα τα ε, σιδηροδρομικά και συμφωνώ με το Street, Ποτέ δεν έχω δει τα έξι σημαντικότερα σχέδια να ήταν σιδηρόδρομοι στα κράτη-μέλη, κυρίως ήταν αυτοκινητόδρομοι και καμιά φορά άκουγες και κανένα τρένο. Ε, εμείς σε επίπεδο ευρωπαϊκό και οικολογικό ήμασταν τρομερά πρωτοπόροι. Ε, τελικά όμως ήρθε το Συμβούλιο και η Κομισιόν και είπε αφήστε τα αυτά τέλος. Ε, είναι πολύ χαμηλή η ποσόστοση τώρα της χρηματοδότηση και δεν υπάρχουν κίνητρα για τα κράτη-μέλη να προωθήσουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Έτσι, αυτά θα πρέπει να τα γνωρίζουμε. Ε, ξέρουμε όμως ότι άμα πάμε από 20 δι σε 8 δι δεν το αποφασίσαμε εμεί, αλλά αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Λοιπόν, που άρχισαν να λένε ότι αυτά τα διάφορα διευρωπαϊκά δίκτυα δεν μπορώ να τα χρηματοδοτήσω μόνο μου στο Μόναχο, στη Στουτγκάρδη, δεξιά και αριστερά να τα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μα οι ίδιοι έρχονται και περικόπτουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια πού θα τα βρούμε τα λεφτά ε, θα πρέπει να πούμε πού είναι η ευθύνη κιόλας για αυτά τα ελλείμματα και τι μειώσεις ευχαριστώ Τελευταίο στον πρώτο γύρο για ε, του συντονιστέ, ο κύριο Μπράτμπορν από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Συγκεκριμένα θα περιοριστώ στις γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν στους διάφορους ε, οργανισμούς, agencies. Όσοι ήσασταν ε, και πριν στην Επιτροπή θα ξέρετε ότι δεν είμαι ενθουσιώδης υποστηριχτής των οργανισμών, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν αξίζουν τα λεφτά τα οποία επενδύουμε σε αυτούς ως προς ε, την βιωσιμότητά τους ε, και τον επαγγελματισμό προσφέρουν στον τομέα της ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας. Ε, εδώ προτείνουμε αύξηση των, ε, της ανάληψης υποχρεώσεων για την ΕΑΣΑ χωρίς όμως να γνωρίζουμε αν επιτελεί τα καθήκοντά της ως δι αυτή η υπηρεσία. Τα τελευταία χρόνια από τη συγκρότησή της δηλαδή δεν έχει καταδειχθεί η ικανότητα να επιτελεί αυτά τα καθήκοντα που τις έχουμε αναθέσει. Αφήστε να, τι θα γίνει αν διευρύνει κρίνουμε και τα καθήκοντά της ε, τώρα. Ε, σε σχέση με την τιμολόγηση και την ε, δομή του κόστους μέσα στον οργανισμό, δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι λειτουργικό το σύστημα, οπότε εγώ στην εκλογική μου περιφέρεια παίρνω καταγγελίες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα, γιατί συνεχώς καλούνται να καταβάλουν μεγαλύτερο κόστος για την πιστοποίηση μικρών, πολύ μικρών τεχνικών προσαρμογών σε ελαφριά μικρά αεροσκάφη. Δεκαπλάσια είναι το κόστος που καλούνται να πληρώσουν. Οπότε εμεί τι κάνουμε, πώ αντιδρούμε, λέμε α δώσουμε περισσότερα κονδύλια. Στο παρελθόν, στην Επιτροπή μα και στο Κοινοβούλιο, για του τέτοιου οργανισμού, τελικά επιπρόσθετα πόσα μπαίνουν σε ένα απόθεμα μέχρι να καταδειχθεί ότι ε, είναι αποτελεσματικός ο οργανισμός. Αυτό πρέπει να κάνουμε γιατί κατά τη γνώμη μου έχει αποτύχει αυτός ο οργανισμός οπότε θα δημιουργηθούν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα αν αυξήσουμε τη χρηματοδότηση τελικά. Ωραία, έχω ακόμα. Έχω ακόμα πέντε ομιλητές και θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών γιατί θα ήθελα να προχωρήσουμε με την έκθεση Γιάνσεν πριν φτάσει και η συγγραφεύς ε, της εκθέσεως, ο κύριος Κόκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το τρίτο πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια λύγει και έχουμε το μεγάλο, είχαμε μεγάλο στόχο συγγνώμη, που δεν φτάσαμε σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό χρειάζεται και ένα τέταρτο πρόγραμμα με χρηματοδότηση ε, ξέρω ότι δεν είναι το πάνω, αλλά χρειάζεται έρευνα, πιλωτικά προγράμματα και για την επιμελητεία και για τις υποδομές. Γι' αυτό ζητώ την απαραίτητη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιάννα Σέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, πρώτον, συμφωνώ απολύτως με τη, το συμπέρασμα του κυρίου Κόχλιτσεκ που απορρίπτει όλες τις περικοπές του Συμβουλίου και ακόμα περισσότερο σήμερα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα των διευρωπαϊκών δικτύων. Το ακριβώς εμείς γνωρίζουμε και ζητήσαμε να πούμε πόσο σημαντικό είναι στο σχέδιο της ανάκαμψης της οικονομίας από όπου είχαν εξεφανιστεί και για την εκτελεστική υπηρεσία για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τον οργανισμό και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να μας ε, πει που βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τον Μάρκο Πόλο λυπάμαι πάρα πολύ. Θα μπορούσε ο κύριος Καραμίτσος να μας εξηγήσει με ποιον τρόπο ε, προτίθενται να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόγραμμα που υποτίθεται ότι είναι του μέλλοντος και ποντάρουμε σε αυτό όπως είναι η δια των ε, μεταφορών και οι λεγόμενοι ε, αυτοκινητόδρομοι λεωφόροι στη θάλασσα. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί αυτό το θέμα δεν μπορεί να ξεκινήσει να απογειωθεί. Και για τα πιλωτικά προγράμματα, συμφωνώ απολύτω με αυτά που είπατε για την οδική ασφάλεια. Θα ήθελα και ο Σκόχλητσέκ να μπει λίγο περισσότερο στην ουσία των πιλωτικών προγραμμάτων για τον τουρισμό που τώρα ξεκινάνε. Και θα ήθελα επίσης να θυμίσω στον πρόεδρο της Επιτροπής μας, τον κύριο Σίμψον, ότι εχθές κάποια στιγμή θυμήθηκα ότι σε καμία περίπτωση αυτή η Επιτροπή που επιγράφεται ε, μεταφορών και τουρισμού δεν συζητάει ποτέ θέματα τουρισμού. Ε, κάποια στιγμή θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τον τουρισμό παρόλο που γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος φόρτος ε, νομοθετικός αλλού, αλλά στο μέλλον θα υπάρχει νομοθετική βάση και θα πρέπει να επικεντρωθούμε και σε αυτό. Και αν μπορούσε ο κύριος Κόχλιτσεκ να πει και τίποτα παραπάνω για τα πιλωτικά προγράμματα του τουρισμού. Τώρα για την ΕΑΣΑ, ίσως θα πρέπει να μας εξηγήσει καλύτερη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι είναι το αντικείμενό τη, σε πάση περιπτώσει, γιατί στην Ισπανία έγινε κάποια παρεξήγηση για το ποιο είναι το αντικείμενο, ποια είναι η αποστολή, γιατί σε ορισμένα ατυχήματα συμμετείχε ε, στη διερεύνηση κάπως αποσπασματικά, αλλού υπάρχουν προβλήματα. Να μάθουμε γιατί υπάρχουν εκεί δυσκολίες και δυσλειτουργίε, υπάρχει έλλειψη προσωπικού ή τίποτα άλλο. Και για την έμψα, για την ασφάλεια στη θάλασσα, γιατί εκτοξεύεται η ανάληψη υποχρεώσεων και ε, περιορίζονται πληρωμέ. Οι εξηγήσει και πάλι δεν με ικανοποιούν. ίσως θα μπορούσε ο κ. Καραμίτσο να μα εξηγήσει πού οφείλονται όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Uh, πολύ ωραία. Μπορώ βέβαια να διαβεβαιώσω όλα τα μέλη ότι ο πρόεδρός σας ε, ε, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιος είναι το της Επιτροπής και με τι πρέπει να ασχολείται. Η κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια ε, γιατί ανήλθατε πλέον και είστε πρόεδρος της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια ε, σχετικά με την αύξηση των κονδυλίων για την ΕΑΣΑ. Ε, κοιτάξτε, ενδεχομένως είναι πολύ αυτό που θα πω και όχι σωστό, αλλά Κάτι που θέλω να πω είναι και ακολουθώ τη σκέψη του συναδέλφου Μπάτμπορν. Είναι ότι θα πρέπει τελικά να αποφασίσουμε εάν η Άσα είναι μια ανεξάρτητη αρχή ε, η οποία δεν στηρίζεται οικονομικά στους κατασκευαστές ή εάν είναι περισσότερο μια ε, ε, υπηρεσία η οποία ασχολείται με την ασφάλεια, γιατί θεωρητικώς αυτό θα έπρεπε να είναι γιατί πιστεύω ότι οτιδήποτε σχετίζεται με το προϋπολογισμό θα πρέπει να λάβει υπόψη το αντικείμενο της ε, υπηρεσίας αυτής, του φορέα αυτού. Φαίνεται ότι οι κατασκευαστές στην ε, Ευρώπη ε, έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει και η FIA που είναι μια υπηρεσία την οποία θα πρέπει να στηρίξουμε γιατί δουλεύει σε όλο τον κόσμο. Απόψή μου είναι ότι όσο τουλάχιστον περνάει ο λόγος μας κύριε Πρόεδρε στην Επιτροπή εδώ θα πρέπει να, έχουμε, να οργανώσουμε μια συζήτηση εγώ δεν λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή το Κοινοβούλιο θα είναι αυτή που θα δίνει όλα τα χρήματα σε αυτές τις υπηρεσίες, αλλά ε, θα πρέπει να αποφασίσουμε εάν πρόκειται να τους επιφορτήσουμε με επιπλέον καθήκοντα, θα πρέπει να προετοιμάσουμε το έδαφος έτσι ώστε τα καθήκοντα αυτά να ληφθούν υπόψη με ικανοποιητικό τρόπο. Απ' την άλλη πλευρά πρέπει να πω ότι οι κατασκευαστές και οι μικροί κατασκευαστές περισσότερο είχαν, αντιμετώπισαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα τον τελευταίο καιρό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, τρεις ε, ομιλητές έχω ακόμα. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα θέλω να πω μόνο για το πώς δικαιολογούνται τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Από ό,τι φαίνεται, το επιχείρημα για τη συγκοινωνία και τις μεταφορές φαίνεται να έχει εξαντληθεί. Ακούμε συνέχεια για την οικονομία και τη συγκυρία. Αν θέλετε για τη συγκυρία να φτιάξουμε και πυραμίδες. Εκεί να δείτε δουλειά που θα έχει η οικοδομή. Είτε έχει νόημα για τις μεταφορές, είτε δεν έχει νόημα, τότε δεν είναι διευρωπαϊκό, ε, οπότε να το αφήσουμε. Όχι για να φτιάξουμε θέσεις απασχόλησης, αλλιώς να δούμε πώς θα ε, επενδύσουμε στην οικοδομή ή στη θερμομόνωση των κτηρίων μας. Ένα άλλο. Ε, γιατί δεν απορροφώνουν τα κονδύλια. Ε, δεν υπάρχει δυνατότητα στα κράτη-μέλη χρηματοδότηση, Γι' αυτό δεν είναι ότι είναι τεχνητό το έλλειμμα ή το έλλειμμα που αισθανόμαστε απλώς. το θέμα δεν είναι το αισθητό έλλειμμα, αλλά είναι το πρόβλημα ότι υπάρχουν πολλά έργα τα οποία θα επιθυμούσαν τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτηθούν, αλλά δεν μπορούν οι ίδιοι να τα χρηματοδοτήσουν. Ε, αφού δεν ε, πληρούνται τα κριτήρια, καλπάζουμε προς το επόμενο σκάνδαλο. Και δεν μπορώ να το δεχτώ. Για τον Μάρκο Πόλο θα πρέπει να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τα κριτήρια. Γιατί εάν ένα τόσο θετικό πρόβλημα δεν βρίσκει καμία ανταπόκριση, ε, κάπου υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα. Και είμαστε υποχρεωμένοι να το λύσουμε. Και μάλιστα τώρα, βραχυπρόθεσμα. Τώρα, για τον τουρισμό, συμφωνώ. Βεβαίω θα πρέπει να κάνουμε συζητήσει. Για παράδειγμα, προτείνω να γίνει μια συζήτηση για αυτό που είχαμε και στην Ολομέλεια τις προάλλε, για αυτή την ιστορία με την Ισπανία και τις ε, κατοικίες ε, της ε, εξοχικές. Θυμάστε έγινε μια μεγάλη φασαρία στην Ολομέλεια, καλό θα ήταν να το συζητήσουμε και Επίσης, ξέρετε, αυτό το θέμα δεν είναι μόνο ισπανικό, απαντά και σε άλλα κρατημέλη και επειδή είναι γενικά ε, προβληματικό στον τουρισμό και για την ασφάλεια ε, στις αερομεταφορές το συντομότερο να συζητήσουμε για τις μαύρες λίστες και για τη χρηματοδότηση. Μήπως αυτό θα έχει ήδη επιπτώσεις ή έχει επιπτώσεις στον προπολογισμό αργότερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκράντες Πασκουάλ. Ανάποδα σας το είπα <laughs> το, το όνομά σας προηγουμένως, ζητώ συγγνώμη. Σας είχα πει Πασκουάλ Γκράντες. Ευχαριστώ κύριε Σίμψον. Συγχαρητήρια για τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνετε. Είμαστε βέβαιοι ότι θα τα ασκήσετε πάντα με ισορροπία και τη συμπάθεια που σας χαρακτηρίζει και πάντα δείχνετε εδώ. Δύο σύντομα σχόλια. Και τα δύο είναι επικρίσεις. Όχι για εσά προφανώς, αλλά Πρώτον, καθυστέρηση στις προπαρασκευαστικές εργασίες διαφόρων ε, σχεδίων προτεραιότητας. Πιστεύω ότι στη θητή αυτή εμείς θα πρέπει να είμαστε απαιτητικοί. Μετά τις μεγάλες εκπτώσεις που είδαμε και έχουμε ένα τσεκούρωμα στον προπολογισμό, 8 δις, ε, είναι απαραίτητο αυτά τα, τα έργα προτεραιότητας να ακολουθήσουν με αντίστοιχο ρυθμό παρά την έκπτωση αυτή για να ευοδοθούν. Είναι λυπηρό το σχέδιο υπαριθμών 7 ο άξονας αυτός συνδυασμένων μεταφορών Πορτογαλία, Ισπανία, Κεντρική Ευρώπη το 2010 είναι ελληματικός από πλευράς χρηματοδότησης. Αυτό είναι απαράδεικτο και θα πρέπει να το καταδικάσουμε. Τώρα για την ΕΜΣΑ, για την ασφάλεια στην αυσιπλοεία και εγώ λυπάμαι για ε, τις περικοπές πιστός πληρωμών εγώ διατέλεσα εισηγητή του κανονισμού για τη χρηματοδότηση του πολιετού κανονισμού για την υπηρεσία αυτή και είχαμε προβλέψει ε, ρυθμίσεις για να μην έχουμε τέτοια καθυστέρηση. Μπορεί η ίδια υπηρεσία να ε, εκτελεί τον προπολογισμό της αποτελεσματικά και στον τύπο και στην ουσία και εγκαίρως. Γιατί έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Κανονικά δεν θα πρέπει να είχαμε τέτοιες καθυστερήσεις. Αυτά, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τικάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ασχοληθώ λίγο με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Δυστυχώς έχουν αργοπορήσει πάρα πολύ τα σχέδια αυτά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε κάνει μάλιστα μία έκθεση η οποία κατεδείκνυε ότι λόγω αυτών των καθυστερήσεων ακριβώς ε, έχουν σπαταληθεί πάρα πολλά χρήματα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρξει αύξηση του κόστους της εφαρμογής των διευρωπαϊκών δικτύων. Θα ήθελα να δούμε το θέμα αυτό από ευρύτερη οπτική γωνία, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την μελλοντική διεύρυνση των διευρωπαϊκών δικτύων. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα έχει συζήτηση επί της αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό των ε, προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από τον επόμενο προϋπολογισμό. Ε, από τη στιγμή που εδώ ενέχονται και τα πιλωτικά προγράμματα και όλη η προπαρασκευαστική εργασία που έχουμε κάνει, ε, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα αρνητική αυτή η μείωση των κονδυλίων. Πιστεύουμε ότι πολλά θα χάσουμε ε, με την κίνηση αυτή, γιατί αντιθέτως από ό,τι συνέβη, εμείς ζητούμε αύξηση των ε, κονδυλίων. Πολλά πρέπει να οικοδομηθούν ακόμα. Δυστυχώς βλέποντας αυτό το προσχέδιο του προϋπολογισμού διαπιστώνουμε μείωση των ποσών αντί για αύξηση. Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές είναι γεγονός ότι το Μάρκο Πόλο θα πρέπει να ε, προωθηθεί περισπεραιτέρω. Θα πρέπει οπωσδήποτε οι εσωτερικές ε, μεταφορές των εσωτερικών δηλαδή πρωτών και οι θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει πρέπει ε, να προωθηθούν περαιτέρω. Ο Δούναβης επίσης θα πρέπει ε, να αποτελέσει κεντρικό σημείο της πολιτικής μας και προτείνω σύσταση ε, ενός intergroup για την κατάσταση στο Δούναβη. Ε, σχετικά με τους ε, ιδιαίτερης αξίας τουριστικούς προορισμούς βλέπουμε ότι και σε αυτό ο προϋπολογισμός δεν κάνει καμιά προσπάθεια να αυξήσει τα κονδύλια. Πρόεδρος, ευχαριστώ Σιλβία. Ο κύριος Πακέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κύριος Ρότερ. Okay. <laughs> Uh, uh, um, Κύριε Πρόεδρε, ήρθα νωρίτερα και δυστυχώς πρέπει να πληρώσω το τίμημα γι' αυτό. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σα συγχαρώ για την ε, ε, ανάληψη της Προεδρίας. Θα μιλήσω για την πολιτική μεταφορά μετά, αλλά θα ήθελα να σχολιάσω μερικά από τα θέματα που ακούστηκαν μέχρι τώρα και οι άλλοι μου συνάδελφοι θα απαντήσουν λεπτομερώς για θέματα τα οποία ε, είναι της αρμοδιότητάς τους. Δυστυχώς αυτός που είναι υπεύθυνος για τον προπολογισμό δεν είναι εδώ. Λοιπόν, να σας πω μερικά πληροφοριακά στοιχεία. Πέρσι δουλέψαμε από κοντά μαζί έτσι ώστε να γίνει το Μάρκο Πόλο ένα επιτυχημένο πρόγραμμα. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι έχει αναλυφθεί πολύ, έχουν αναλυφθεί πολύ ορθότερες ε, ε, προοπτικές για το Μάρκο Πόλο από ό,τι στο παρελθόν. Στο παρελθόν δεν δούλεψε καλά το πρόγραμμα Μάρκο Πόλο, αλλά τώρα σιγά σιγά οδεύουμε προς μια κατάσταση όπου το πρόγραμμα είναι καλό αλλά δεν έχουμε αρκετά χρήματα. Αυτή είναι λοιπόν μια πρώτη πληροφόρηση και μετά ε, θα μιλήσω αργότερα εν λεπτομερία. Ε, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε επίσης και στην Executive Agency. Έγινε πολύ καλύτερο το πρόγραμμα, εξήγησε πολύ καλύτερα πώς μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερα στο πρόγραμμα αυτό όσον αφορά όσον αφορά ε, την ε, χρηματοδότηση των ε, διευρωπαϊκών δικτύων. Ξέρει πολύ καλά το Κοινοβούλιο πώς είναι τα πράγματα και βεβαίως δεν χρειάζεται να πω ότι λυπούμε και εγώ για την περικοπή των κονδυλίων, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να πορευτούμε με τον προπολογισμό που έχουμε τώρα. Αργότερα θα αναφερθώ ε, και στο πρόγραμμα οικονομικής ε, ανάκαψης ε, και τα 500 εκατομμύρια τα οποία, με τα οποία θα επαναχρηματοδοτήσουμε τον προϋπολογισμό όσον αφορά... Όσον αφορά την ΕΑΣΑ δεν θα πω στην ουσία του πράγματος. Νομίζω πάντως ότι θα πρέπει να έχουμε περαιτέρω συζήτηση για την ΕΑΣΑ. Πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστές φιλοσοφίες. Δηλαδή Έχουμε ρυθμιστική υπηρεσία η οποία ασχολείται με την ασφάλεια ή έχουμε και η οποία ε, έχει ε, δημόσια χρηματοδότηση ή έχουμε μια άλλου είδους υπηρεσία η οποία βασίζεται σε τέλη ε, κλπ. Εδώ νομίζω ότι έχουμε ένα, μια ανάμιξη ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης αλλά πρέπει να επανέλθω σε αυτό. Η κυρία Γιάλα αναφέρθηκε στο θέμα της ε, διερεύνησης ατυχημάτων. Νομίζω ότι ε, όταν θα αναφερθώ στις μελλοντικές πολιτικές της Γενικής μας ε, Διεύθυνσης θα έχει απάντηση στα ερωτήματά της όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Ακόμα ένα θέμα, αυτό που ανέφερε η κυρία Τικάου, θα ήθελα να αναφέρω. Κοιτάξτε, εμείς ε, ασχολούμαστε πολύ σε όλα τα αρμόδια τμήματα της Επιτροπής ε, στο, για το θέμα του Δούναβη. Έχουμε αυτή τη στιγμή και έναν συντονιστή για την αυσιπλοεία των εσωτερικών πλωτών οδών αλλά παρόλα αυτά ε, καταγράφω το σημείο το οποίο ανέφερε και στους επόμενους μήνες οπωσδήποτε ε, θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε μία πιο στοχευμένη και συνολική πολιτική για το Δούναβι όπως κάναμε για την ε, Βαλτική και για κάποιες άλλες περιοχές. Αυτά ήθελα να πω για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ρόιτε, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι όλοι αγαπάμε τον Δούναβη και χαίρομαι που θίξατε και το θέμα του Δούναβη. Χρονοδιάγραμμα λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Α, θέλεις να πεις κάτι άλλο. Ναι. Ε, ε, ναι, Μπράιαν, θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ο κύριος Πακέ σε σχέση με τον προπολογισμό των διευρωπαϊκών δικτύων. αυτό που βάλαμε για το σχέδιο ανάκαμψης οικονομίας για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Μήπως μπορεί να μας δώσει καμία λεπτομέρεια παραπάνω, αν γίνεται. Λοιπόν, ναι, ναι, θα γίνει μετά αυτό. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών 14, 14 Αυγούστου. Ακριβώς στη μέση των διακοπών σας και είμαι βέβαιος ότι όλοι μόνο γι' αυτό θα δουλεύετε, όπου και αν βρισκόσαστε, θα δουλεύετε σκληρά για τον προϋπολογισμό έγκριση στην Επιτροπή Μεταφορών προβλέπεται για, για τη Δευτέρα Σεπτεμβρίου και στην Ολομέλεια τον Οκτώβρη, ε, Σύνοδο Ολομελίας του Οκτωβρίου. Θα το ξανασυζητήσουμε στη δεύτερη συνάντησή μας του Σεπτεμβρίου και μετά στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Θα κάνουμε λοιπόν πρώτη συζήτηση, πρώτη ανταλλαγή απόψεων 2 Σεπτεμβρίου, ε, δεύτερη συζήτηση στη δεύτερη συνάντηση του Σεπτεμβρίου και στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου θα φτάσει το θέμα αυτό. Θα ήθελα να πω σε όσους ένθιξαν το θέμα αυτό. Εμείς καλέ, ότι καλέσαμε τον κύριο Μπουντρών της ΕΑΣΑ στην ενάντησή μας, στην ιδρύασή μας του Σεπτεμβρίου και επομένως μπορείτε τότε να του υποβάλλετε όλα τα σχετικά ερωτήματα, τα οποία φαντάζομαι θα είναι πολυπληθή. Πολύ ωραία. Επόμενο σημείο είναι τα ITS. Η κυρία Γένσεν, παρακαλώ. Jeg skal fortælle lidt om, hvor vi er henne med ITS-handlingsplanen. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα σας πω που έχουμε φτάσει λοιπόν με τα προγράμματα αυτά. Τα ευφύ e συστήματα μεταφορών λοιπόν, ITS, που αφορά μια σειρά διαφορετικών πραγμάτων. Ε, δηλαδή πηγαίνει από, τον, ε, ε, από συστήματα επικοινωνίας δεν έχει τίποτα. Από συστήματα, λέω, παρακολούθησης ε, μέχρι ε, καινούριες ε, τεχνολογίες στις οδικές μεταφορές. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε την διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στα διάφορα είδη μεταφορών. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε στα τέλη του 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο κάναμε μια πρώτη εξέταση του ζητήματος και μάλιστα το εγκρίναμε και στην Ολομέλεια. Όμως υπάρχουν δύο σκέλη τα οποία συνδέονται. Ε, πρώτα απ' όλα όσον αφορά την προσέγγιση της Επιτροπής, ε, αυτή έχει απομονώσει έξι διαφορετικούς ε, ε, ε, διαφορετικά πεδία επί των οποίων ε, θα πρέπει να κινηθεί ας πούμε τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να δίνονται στους οδηγούς άρα ένας σύσταση καταλόγων στοιχείων επίσης κατάρτιση καταλόγου σχετικά με τις, ε, ε, τους εξοπλισμούς ασφαλείας, τον τρόπο με τον οποίο ε, οι εξοπλισμοί αυτοί αποθηκεύονται. Μία σειρά από δεδομένα. Απ' την άλλη πλευρά, η θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την πρωτοβουλία της Επιτροπής είναι ότι δεν θεωρούσαμε ότι υπήρχε λόγος να υπάρξει οδηγία γιατί δεν χρειαζόταν κάτι τέτοιο έτσι ώστε ε, το έτσι ώστε τα κράτη-μέλη ε, να είναι υποχρεωμένα ε, να ακολουθήσουν αυτές τις δεσμευτικές διατάξεις. Και φαίνεται ότι εκεί υπήρξε μια διαδικασία αμφισβήτησης ανάμεσα στην Κομισιόν και το Συμβούλιο για το βαθμό δεσμευτικότητας που θα έχουν τα μέτρα αυτά. Ε, βέβαια πρέπει να γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε αυτό το σύστημα ε, των ευφυών συστημάτων μεταφορών θα πρέπει κάποια στιγμή να κινηθούν ε, γιατί εδώ αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου ο ένας στέλνει τον μπαλάκι στον άλλον και αναρωτιόμαστε αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα λέει η ομιλήτρια. Ε, βεβαίως το ζήτημα είναι, ε, συμφωνούμε όλοι για τον εξοπλισμό που θα πρέπει να ε, υπάρχει, αλλά δεν συμφωνούν ας πούμε αν θα πρέπει ο εξοπλισμός αυτός να είναι ε, συνδεδεμένος με το όχημα και πώς θα πρέπει να, θα πρέπει να είναι δεσμευτικός, υποχρεωτικός ο εξοπλισμός αυτός και πρέπει να είμαστε, ε, να συμφωνήσουμε ε, πάνω σε ορισμένα θέματα. Επομένως, το action plan ε, και η οδηγία ε, έχουν αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας. Όμως, ε, όλος ο σκοπός ο οποίος βρίσκεται πίσω από το σχέδιο δράσης ακόμα δεν είναι σαφής. Πάντως, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ανταλλαγή εμπειριών, τις οποίες θα μελετήσουμε, έτσι ώστε να δούμε με ποιο τρόπο και ποιου είδους στάνταρ θα πρέπει να καθορίσουμε και τον τρόπο βεβαίως που θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Η αρχική προσπάθεια ήταν να συμφωνήσουμε πάνω στα, στις στα πεδία αυτά ε, για τα οποία, για τα στάνταρ μάλλον των οποίων, τα πρότυπα των οποίων μπορούμε να συμφωνήσουμε ε, και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Από την άλλη πλευρά βεβαίως εμείς δεν θέλουμε να υπογράψουμε λευκή επιταγή στην Επιτροπή ε, η οποία επιτροπή με τη σειρά της ε, θα αποφασίσει και θα επιβάλλει στα κράτη-μέλη ε, ό,τι της περάσει από το κεφάλι. Άρα χρειαζόμαστε κάποια σαφήνεια εδώ. Ε, θέλουμε καθαρότητα των θέσεων της Επιτροπής από την άλλη πλευρά. Θέλουμε να ξέρουμε πόσο θα κοστίσει όλο αυτό το εγχείρημα. Γιατί όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά, αλλά θα πρέπει να τα δούμε συνολικά ε, και δεν είναι δυνατόν ε, να υποχρεώσουμε από την αρχή όλα τα κράτη-μέλη ε, να κάνουν, να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Μπορούμε να προχωρήσουμε πρώτα απ' όλα με ένα μνημόνιο συνεργασίας και η Τσεχική, Δημοκρα... η Προεδρία συγγνώμη, και η Σουηδική Προεδρία τώρα φαίνεται ότι θέλει να ασχοληθεί με τα ευφύ συστήματα μεταφορών έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια σειρά κοινών κανόνων, τουλάχιστον σε ορισμένα πεδία, ενώ, το, οι οποίοι θα είναι δεσμευτικοί. Ενώ σε κάποια άλλα πεδία μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ε, θα καταρτήσουμε μια σειρά κανόνων ε, που ε, δεν θα είναι δεσμευτικοί και υποχρεωτικά εφαρμόσιμοι από τα κράτη-μέλη. Και βεβαίως επί τη βάση όλων όσων έχουμε δεχτεί και στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου μπορούμε να ξεκινήσουμε σε άτυπες συζητήσεις με το Συμβούλιο. Αυτό που θα ήθελε η Σουηδική Προεδρία είναι να επιτύχει μία πρώιμη συμφωνία ε, στην φάση της πρώτης ανάγνωσης. Μία συμφωνία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα περάσουμε εύκολα ε, στην πρώτη ανάγνωση. Δεν ξέρω βεβαίως πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό ως προσέγγιση μπορούμε να το συζητήσουμε και στους ε, συντονιστές και θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα στόχο για μας γιατί αυτές οι διαπραγματεύσεις ε, πράγματι θα μπορούσαν να γίνουν από μένα ε, και από τους σκιώδεις των άλλων ομάδων και να δώσουμε το απαραίτητο feedback στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής και με τον τρόπο αυτό ε, θα ε, επιβεβαιώναμε ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε την γραμμή που ενέκρινε το προηγούμενο κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, θα το συζητήσουν οι συντονιστές. Φυσικά. Και για την υπόλοιπη νομοθεσία που έχει να κάνει με την πρώτη ανάγνωση. να δούμε πώς θα γίνει η δεκτή αυτή και πώς θα προχωρήσουμε. Μετά τη συνεδρίαση θα το συζητήσουν οι συντονιστές και θα έχετε απάντηση. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Γκρός από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ja, genau, wollte kurz zur Prozedur. Ich bin kein... Ε, σύντομα, ε, διαδικαστικά. Δεν είμαι σχολαστικός εγώ και ψήρας εντός εισαγωγικών, αλλά καλό είναι να πούμε εδώ στην Επιτροπή και για τους συναδέλφους τι γίνεται με τις εκθέσεις που ολοκληρώνονται σε πρώτη ανάγνωση. Αυτές οι εκθέσεις εγκρίνονται ως έχουν και μετά ε, εμείς εδώ στην Επιτροπή μας συνεχίζουμε να τις συζητάμε. Η κυρία Γιάννησεν το ζήτησε και μπήκε στην ημερήσια διάταξη και μπορεί ενδεχομένως να προχωρήσουμε ε, σε πρώιμη ε, συμφωνία. Αυτό τι σημαίνει το early agreement, ότι θεωρούμε ότι θα λυθεί σε πρώτη ανάγνωση και ήδη από σήμερα θα πρέπει να λάβουμε απόφαση, τέτοια πρόθεση έχετε, γιατί θα πρέπει να ορίσουμε και σκιώδεις ηγητές οι πολιτικές ομάδες και ε, να συνεργαστούμε και με τη Σουηδική Προεδρία. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις για να μπορέσουν να συμμετέχουν και οι σκιώδεις ηγητές. Αυτό ήταν το διαδικαστικό. Προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα και γενικά θα συμφωνούσα αν ισχύσει το ίδιο που ισχύει και στις άλλες εκθέσεις ε, που ολοκληρώνονται σε πρώτη ανάγνωση. Τώρα, επί της ουσίας, θεωρώ ότι στην Επιτροπή μας εδώ το υποστηρίξαμε σχετικά μεγάλη πλειοψηφία όλο αυτό το εγχείρημα. Γνωρίζουμε τις επιφυλάξεις και του Συμβουλίου. Είναι γενικές οι επιφυλάξεις που έχουν στο Συμβούλιο, όχι μόνο για αυτό το θέμα. Πάντω, γενικά μπορούμε να πούμε ότι εδώ για τη σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή πρώτον για να προωθηθεί η ασφάλεια και αυτό θα πρέπει να μείνει με το οποίο να εκπέμπουμε και προ τα έξω και το δεύτερο αυτό που όπως πολύ ωραία ονομάζεται ΕΦΕΙΣ μέθοδοι μεταφορών ε, να οδηγήσουν και στην προστασία του περιβάλλοντος και σε αντίστοιχα μέτρα με στοιχεία και ημερομηνίε ε, που αναφέρονται εδώ. Και το τρίτο, για την προστασία των δεδομένων, πιστεύω ότι η κατάσταση που όπως έχει ε, σήμερα χρειάζεται συντονισμό στα διάφορα κράτη-μέλη. Προς το παρόν επικεντρώνονται στα τεχνικά θέματα για να επεκταθούν οι δυνατότητες τεχνολογικές που υπάρχουν σήμερα. Κάτι άλλο που είπαμε ήδη και στον προϋπολογισμό. Να υπάρχουν λεγόμενες ασφαλείς θέσεις ε, στάθμευσης για ε, φορτηγά δημόσιας χρήσης και να τα γνωρίζουν και τα συστήματα πλοήγησης και να φαίνονται. Θα πρέπει να ε, γίνει μια μετάβαση τώρα από αυτά που πρεσβεύουμε ε, θεωρητικά και αυτά που μπορούμε να εφαρμόσουμε στην πράξη και από οικονομικής απόψεως. Και αυτό πρέπει να το συνδέσουμε και με τον προπολογισμό αλλά και με τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης όπου γνωρίζουμε ε, πολύ καλά ότι στις ζωτικές μεταφορές υπάρχουν πολλά προβλήματα διότι δεν υπάρχουν ασφαλή πάρκινγκ για να μην πω ότι δεν υπάρχουν καθόλου πάρκινγκ. Πού να σταματάνε οι άνθρωποι για να αναπαύονται. Λοιπόν, καλά όλα αυτά να τα λέμε, αλλά λέμε μετά ότι είναι και υποχρεωτικά όλα αυτά που αποφασίζουμε ω κέντρα βάρου και σημαντικά στου διάφορου τομεί να χρηματοδοτούνται και να υλοποιούνται. Χαίρομαι για την ε, προσπάθεια της κυρίας Γένσεν και καλωσορίζω την έκθεση και θα ευχόμουν να προωθηθεί γρήγορα το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας και ελπίζω και η σημερινή Προεδρία να δείξει προθυμία να προχωρήσει στο θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, θα δούμε τι θα προκύψει από τις συνεδρίες... Αν μετά από τη συζήτηση θέλουμε να ε, εγκρίνουμε στην πρώτη ανάγνωση τα 5-6 ντοσιέ αυτά, μέσα στην πρώτη ανάγνωση ξαναλέω, να το προωθήσουμε γιατί θα επισπεύσουμε έτσι τις εργασίες μας. Και έτσι ο εισηγητής ε, που ασχολείται ακόμη με το θέμα θα μπορέσει να συνεχίσει άμα κάνουμε τις απαιτούμενες αλλαγές θα έχει η Επιτροπή το χρόνο να επισπεύσει τη διαδικασία, να διευκολύνει τις αλλαγές. Ε, θα δούμε. Ας τελειώσει πρώτα η συζήτηση. Ο κύριος Λάιχσφριντ. Από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ για τη διαδικασία. Θα υποστήριζα και εγώ αυτή την πρόταση. Τώρα έχω νομίζω Έχουμε εδώ πέντε ή έξι εκθέσεις που είναι έτοιμες, που έχουν ολοκληρωθεί και αποφασιστεί πλήρως. Έξι, ε, έξι είναι, έξι παρακαλώ, έτοιμες εκθέσεις που έχει ολοκληρωθεί η δουλειά στο έτοιμε που κοινοβούλιο και αποφασιστει πληρως εξι ειναι δουλειά ετών πολλές φορές και δεν θα είχε νόημα να ξανανοίξουμε αυτές τις εκθέσεις, να αλλάξουμε οτιδήποτε. Θα ήμουν κι εγώ υπέρ λοιπόν του να το ξεκαθαρίσουμε σήμερα αυτό, να το διεκπαιρεώσουμε και να επιβεβαιώσουμε τις εκθέσεις των συναδέλφων της προηγουμένης περίοδου. Και είναι πιο απλά τα πράγματα για να ξέρουμε τι μελιγενέστε σε όλες τις εκθέσεις. Αν κάποιος θέλει αλλαγές, ακολουθούμε τη συνήθεια διαδικασία. Με ε, τη δυνατότητα υποβολής τροπολογιών σε δεύτερη ανάγνωση και αυτή καλή λίστα ήταν. Ε, και εγώ συμφωνώ με την κυρία Γένσεν. Θα έπρεπε να προσπαθήσουμε τώρα τη συγκεκριμένη αυτή έκθεση να την ολοκληρώσουμε σε μια πρώιμη συμφωνία και σε δεύτερη ανάγνωση και προσφέρονται για τέτοια διαδικασία θέματα που στο Κοινοβούλιο βρίσκουν ευρύτατη συνένεση. Ε, καλά συνεννοούνται οι συγκητριακές και οι Και εγώ το έκανα στη δική μου έκθεση. Χρειάστηκαν δύο χρόνια και αναλώθηκαν τρεις προεδρίες αυτό, αλλά τελικά ευωδόθηκε. Και ελπίζω ε, στην κυρία Γιάννησεν τα πράγματα να πάνε καλύτερα τώρα. Ε, σε ό,τι αφορά την ουσία δεν έχω πολλά να πω. Το εξή μόνο. Δύο πράγματα είναι σημαντικά για μένα. Πρώτον, όσο πιο εντατική είναι η δικτύωση των συμμετεχόντων στις μεταφορές και τις συγκοινωνίες, τόσο μεγαλύτερη είναι και η δυνατότητα ε, να ε, ελέγξει κανείς που πήγαν, πόσες ώρες οδήγησαν, ε, οδηγεί των φορτηγών κτλ. Δηλαδή, για την οδική ασφάλεια και τη ροή ε, της κυκλοφορίας των συγκοινωνιών χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προστασία των δεδομένων γιατί καταγράφονται πολλά δεδομένα και μπορεί κανείς να ελέγχει τα πάντα. Και επίσης τέτοια συστήματα είναι πανάκριβα. Θα πρέπει να φροντίσουμε αυτό να μην επιβαρύνει μόνο τον τελικό χρήστη, Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που κάνουν πολλά χιλιόμετρα για να πάνε στη δουλειά τους, να εργαστούν αλλού, που έτσι και δεν κερδίζουν πολλά χρήματα και δεν θα πρέπει να τα τρώνε όλα στον δρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Greens, Mrs. Από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συστήσω και είναι πολύ σωστό αυτό. Ε, ε, οι εκθέσεις τελευταίας περίοδων έχουν ολοκληρωθεί, να δώσουμε το ok σε όλες τις εκθέσεις για να έχουμε μια καλή βάση, να μην αρχίζουμε από την αρχή την κάθε έκθεση, να μην ξανανοίγουμε τη συζήτηση. Σε περίπτωση που αυτό ισχύει και μπορεί να γίνει, ε, είναι καλό. Τώρα, για την ουσία κι εγώ στο μεταξύ, διάβασα μερικές ενδιαφέρουσες μελέτες. Υπάρχουν μερικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν περισσότερο υπόψη και δεν έχει κυριαρχήσει αυτό στη συζήτηση. Τι έχει διαφανεί. Σε ψυχολογικές μελέτες για τις μεταφορές ξεκάθαρα φαίνεται ότι όσο περισσότερα μέτρα ασφαλείας ε, έχει ενσωματωμένα το αυτοκίνητο, το όχημα, τόσο πιο ρηψοκίνδυνα οδηγεί ο οδηγός. Όταν έχεις ε, ABS, ε, τρέχεις περισσότερο, οδηγείς πιο ρηψοκίνδυνα. Αλλάζει αμέσως η οδική συμπεριφορά και αντισταθμίζει τα θετικά του τεχνικού συστήματος. Οπότε, ερώτηση, είναι σκόπιμο να έχουμε τόσο υψηλή ασφάλεια, χρειάζονται ιδιαίτερα προγράμματα οδικής κατάρτισης και κυκλοφοριακή αγωγή για τους οδηγούς για να ε, οδηγούν λογικά και όχι τρελά. Υπάρχουν και τέτοια θέματα ψυχολογίας οδικής ε, συμπεριφοράς των οδηγών. Πριν υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν δαπάνες ε, αστρονομικές, και όχι μόνο τα κράτη, αλλά και οι μεμονωμένοι οδηγοί. Εάν δεν υπάρχει τελικά ασφάλεια οδική. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και στην προστασία των δεδομένων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πολύ σοβαρά ότι είναι βασική προϋπόθεση και προαπαιτούμενο. Αν δεν το σεβαστούμε αυτό θα αναβαγίσει ολόκληρο το, πρόβλημα, το πρόγραμμα. Και η αντίσταση των κρατών μελών είναι ακριβώς εκεί. Δεν λαμβάνουν καν υπόψη διάφορα θέματα ή τα αγνοούν γιατί είναι πολύ υψηλό το κόστος ή είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η προστασία των δεδομένων. Το έχουμε ξαναδεί αυτά στην έκθεση της συναδέλφου Αγιάλα Σέντερ για τη διασυνοριακή επιβολή των μέτρων αυτών, Ούτε καν την ποινική δίωξη τη διασυνοριακή για βαριά ε, ε, βαριές παραβιάσεις δεν δέχτηκε το Συμβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε για τις τεχνικές υποδομές, να το λάβουμε υπόψη μας, αλλιώς οποιοδήποτε προϋπολογισμός ε, κόστους ωφέλους ή μελέτη αντικτύπου εκτινάζεται και, και, και βγαίνει τελείως εκτός πλαισίου και γίνεται ανέφικτο πραγματικά να κοιτάξουμε τι έχει νόημα, πού ε, είναι σίγουρη η προστασία των δεδομένων, πού εξασφαλίζεται για να λάβουν τα κράτη-μέλη τα μέτρα, να τους πείσουμε δηλαδή εμείς. Ευχαριστούμε. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι τους ευφυείς οδηγούς. Άλλο ενδιαφέρον θέμα. Ωραία, ναι, να μιλήσουμε για τους ευφυείς οδηγούς, λοιπόν. Να αλλάξουμε τον τίτλο. Η κυρία Τικά. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Γένσεν για την παρουσίασή της. Συνεργαστήκαμε αγαστά για το θέμα αυτό, πέραν από την οδική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, εφόσον μιλάμε για ευφυή ε, συστήματα μεταφορών, για τις οδικές μεταφορές αλλά και για τις διεπαφέ, τα interface με άλλα είδη μεταφορών θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το θέμα της αστικής κινητικότητας. Είναι σημαντικό να μην ασχολούμαστε ε, ε, μόνο με τα κονδύλια του προϋπολογισμού των διευρωπαϊκών δικτύων, γιατί επί σειρά ετών σημειώνεται αύξηση στα κονδύλια. Το βλέπουμε αυτό. εδώ και χρόνια και το Συμβούλιο καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο πρέπει να, πρέπει να συζητήσουν τα κράτη-μέλη και να τονιστεί ότι το 2010 θα κάνουμε διάμεση αναθεώρηση σε σχέση με την απορρόφηση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων. Τα διαρθρωτικά κονδύλια είναι επιλέξιμα στο μέτρο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση της αστικής κινητικότητας ε, σε συνδυασμό με τα ευφυή e, συστήματα μεταφορών. Η ομάδα των σοσιαλιστών στο παρελθόν τόνισε την ε, ανάγκη καλύτερης διεπαφής ανάμεσα στα διάφορα είδη μεταφορών και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε βάρος σε αυτήν την ιδέα. Σας ευχαριστούμε για την Επιτροπή. Ο κύριος Καραμίτσος. Ήξερα ότι δεν θα έλεγα καλά το όνομά σα. Εν πάση περιπτώσει, <laughs> κύριο Καραμίτσος. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Ήταν ε, περιεκτική η παρουσίασή της, Παρουσία την τρέχουσα κατάσταση. Ε, χρειαζόμαστε εξελίξεις ε, σε αυτό το τομέα να κάνουμε προσπάθειες ε, ούτω ώστε πρόωρα στο αρχικό στάδιο τη Δεύτερη ανάγνωση, να καταλήξουμε συμφωνία. Βέβαια ε, είναι αφισβητήσιμο το αν θα τα καταφέρουμε. Ένα από τα σημαντικά θέματα ε, είναι ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τις παρελθούσε εργασίες του Κοινοβουλίου. Έχουμε κάνει εκτεταμένες εξωτερικές διαβουλεύσεις, ακροάσει. Έχουμε ακούσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά στην έκθεση που έχει εγκριθεί και υπάρχει νομίζω μια παρανόηση στις επαφές με το Συμβούλιο και προσπαθούμε να την ε, διαλευκάνουμε. Η ιδέα δηλαδή ε, που η φήμη που κυκλοφορεί ότι εμείς θέλουμε επιτα... λευκή επιταγή στην Επιτροπή για να παίρνουμε αποφάσεις. Μα δεν αληθεύει αυτό. Ε, στο, ε, το Συμβούλιο στο Μάρτιο ενέκρινε συμπεράσματα. Εκεί υπάρχουν οι αρχές και οι λεπτομέρειες ε, του σχεδίου δράσης για περιορισμένου, για περιορισμένου αριθμού θέματα. Στη συνέχεια μιλήσαμε για δέσμευση και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι κεντρική σημασία μέσα στην οδηγία. Το ίδιο έχουμε κάνει και για τους σιδηροδρόμους, για τις θαλάσσιες μεταφορές, για τις... Ε, ποτάμιες μεταφορές. Ε, έχουμε την νομοθεσία, προτυποποίηση και στη συνέχεια χρηματοδότηση. Αυτά είναι τα στάδια. Οπότε, εφόσον έχουμε ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση για άλλα είδη μεταφορών, έχουν αναπτυχθεί συστήματα ε, στις ακτογραμμές, στα ποτάμια, στα σημεία σύνδεσης διαφορετικών τρόπων μεταφοράς. Πριν από 10-15 χρόνια είχαμε το το περίφημο ε, σύστημα για ε, τα δεδομένα, για τα αυτοκίνητα, αλλά για να αυξήσουμε την οδική ασφάλεια τώρα και να προστατεύσουμε το περιβάλλον, θα πρέπει να ε, εγκριθούν τα νέα συστήματα, να αρχίσουμε με τις ελάχιστες υπηρεσίες, κατοχυρωμένες υπηρεσίες όπως προτείνει το Κοινοβούλιο, τόσο ώστε να υποφεληθεί και ο κλάδος, η βιομηχανία και να εκπληρωθούν οι στόχοι της πολιτικής μεταφορών. Αυτός είναι ο στόχος των υπό εξέταση προτάσεων, διότι μέχρι στιγμής πρωτοβουλίε ανελήφθησαν μόνο από τον ιδιωτικό τομέα, οπότε χρειαζόμαστε προδιαγραφέ για τις ελαχίστου επίπεδου υπηρεσίε, ούτω ώστε να σημειωθεί γρήγορα πρόοδο και ένα επαγγελματία οδηγό. ή εμείς, άμα θέλουμε να πάμε από τη Στοχόλμη στον Πειραιά, να έχουμε τι ελάχιστες υπηρεσίε, να αποφύγουμε τα ατυχήματα, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και ούτω καθεξής από πλευρά μα. Ε, θέλουμε να συμμετάσχουν ενεργά και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να καταλέξουμε το ταχύτερο δυνατόν συμφωνία. Έχουμε χάσει πάρα πολλά χρόνια, σας είπα 15 χρόνια ε, και θα υποφεληθούμε όλοι τα μάλα. Όχι μόνο οι πολίτες, όχι μόνο αυτοί που εκπονούν πολιτικές, αλλά και η βιομηχανία είναι μια τεράστια αγορά, παγκόσμια αγορά. Πρέπει να καταδείξουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε τους ε, στόχους μας και έτσι θα αποκτήσουμε και περισσότερες επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Άννα, θέλεις να επανέλθεις, θες να κάνεις άλλα σχόλια. Ε, έχω μερικές παρατηρήσεις ακόμα. Εγώ μπορώ να επιβεβαιώσω αυτά που λέγει ο κύριος Καραμίτσος, ότι ε, ουσιαστικά το Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι συμπαραστάτης στην προσπάθεια αυτή είναι δουλειά ετών και επίση ε, έχουμε κάνει ακροάσεις, ομάδες εργασίας. Ε, υπάρχει υλικό ε, το οποίο αποκρισταλώνεται σε αυτή τη τελική θέση και πολύ. Υπάρχει και μια πρακτική αφετηρία. Όταν λέμε θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια παντού στην Ευρώπη, θέλουμε να φροντίσουμε ακριβώς να μην καταλήξουμε στην κατάσταση που έχουμε τώρα. Ξεκινάει ένα φορτηγό από τη Στοχόλμη και πρέπει να πάει μέχρι την Ελλάδα. Πρέπει να κολλήσει ε, περίπου στο Παμπρίστου διάφορα σημειώματα και στίκερ για να ξέρει ο οδηγός σε κάθε χώρα τι ισχύει. Και χάνεται και θα πρέπει να έχει μία μονάδα on-board unit για να καταλαβαίνει και σε γλώσσα που καταλαβαίνει τι ισχύει σε όλη την Ευρώπη και να μπορεί να προχωρήσει. Και το θέμα αυτό που είπε ο κύριος Γκρός για ασφαλείς θέσεις στάθμευσης, τα είπε και η κυρία Τσικάου αυτά. Θα πρέπει ε, να προωθηθεί αυτό το θέμα. Το έχει πιέσει πάρα πολύ η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο και υπάρχει ένα σύστημα για να ταυτοποιηθούν αυτές οι θέσεις πάρκινγκ. Ε, το θέμα είναι ότι δεν εφευρίσκουμε συνέχεια νέα πράγματα, να καταγράψουμε και την πραγματικότητα. Θα πρέπει να ξέρει ο οδηγό που είναι το επόμενο πάρκινγκ, να πάει να σταθμεύσει, να ξεκουραστεί, να μην είναι μέσα στο άγχο να ψάχνει πού θα σταματήσει να αναπαυθεί, να γνωρίζει ε, και να προγραμματίσει του χρόνου οδήγηση, του χρόνου ανάπαυση ε, με σύστημα και με τι σωστέ συνθήκε. Αυτό θέλει και το Κοινοβούλιο. Να είναι καλέ οι συνθήκε διαβίωση και εργασία και απασχόληση των εργαζομένων μεταφορέ. Και ελπίζω να προχωρήσουμε θα ήθελα πέρα από την τεχνολογία και την οικολογία να τονίσω πόσο σημαντικό είναι το θέμα της ασφάλειας. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε ε, ένας οδηγός να μην ε, έχει το πρόβλημα της, ε, να, ε, να μην αποσπάται η προσοχή του την ώρα που οδηγεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οδική ασφάλεια. Και βεβαίω θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μα ότι το πρόβλημα του, του οδηγού, έστω και με τις νέες τεχνολογίες, μπορεί να είναι πάρα πολύ σοβαρό. Επομένω, εγώ είμαι κατά. Ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι διαβλέπετε συνένεση από όλου ότι θέλετε να προχωρήσουμε σε αυτά τα έξι ε, τα, τους έξι φακέλους των οποίων έχει ολοκληρωθεί η πρώτη ανάγνωση. Βλέπω τους ε, έξι συναδέλφους και στρέφουμε προς αυτούς ε, προς επιβεβαίωση ότι μπορούμε να δεχτούμε ε, για πρώτη ανάγνωση και να προχωρήσουμε και βεβαίως αυτό μας δίνει και τη δυνατότητα να ορίσουμε εισηγητές οποτεδήποτε ε, χρειάζεται αυτό και αν δεν έχουμε τους παλιούς εισηγητές. Συμφωνείτε όλοι? Μήπως θα μπορείτε να μου πείτε, να μου δείξετε διανατάσεις της χειρός υπέρ, κατά, αποχές Ντέρκ, δεν απέχει. Θες να πει κάτι. Ναι, Πρόεδρε. Θα διευρύνουμε και τη δυνατότητα για τροπολογίες. Όχι. Αυτό θα ε, ε, σε αυτό θα εφαρμοστεί ο νέος κανόνα σε σχέση και με τη δεύτερη ανάγνωση. Λοιπόν, είπαμε ότι η δυνατότητά σας να υποβάλλετε τροπολογίες βάσει του νέου κανονισμού είναι ε, πολύ περιορισμένος όμως με τον, ε, συγγνώμη, βάσει του παλιού κανονισμού. Βάσει του νέου κανονισμού όμως λέμε ότι όταν δεχτούμε την πρώτη ανάγνωση μπορούμε να προχωρήσουμε σε δεύτερη ανάγνωση αφενός, αλλά ανοίγουμε και τη δυνατότητα υποβολής τροπολογιών εάν κάτι τέτοιο επιθυμείτε. Αν θυμάμαι καλά είναι ο κανονισμός υπαριθμών 7. Δεν είμαι και σίγουρος λέει ο πρόεδρος. Θα το δούμε. Μαθιού. Ναι. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους έτσι με τρόπο έμεσο ότι ε, όλες οι τροπολογίες μπορούν να κατατεθούν αλλά στην Ολομέλεια ε, ψηφίζεται ε, σε δεύτερη ανάγνωση. Δηλαδή, ε, δεν μπορούν να περάσουν με απλή πλειοψηφία αυτές οι τροπολογίες, έτσι. Ήθελα να το πω αυτό για να το ξέρουν οι συνάδελφοι. Μην νομίζω ότι θα κάνουν τροπολογίες και με απλή πλειοψηφία περνάνε. Όχι. Μάλιστα. Ναι. Είναι δεύτερη ανάγνωση, χρειάζεται ειδική πλειοψηφία κτλ. Αλλά μπορείτε να κάνετε τροπολογίες έτσι και έτσι. Κάτι λέει η κυρία Αγιάλα εκτός Μητροφων. Δεν ακούμε. Λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Ανταλλαγή απόψεων με το Γενικό Διευθυντή ε, Τρέν, του κυρίου Μάτιου ε, Ρόιτερ. Μπορεί να έρθει εδώ επάνω και όλοι θα κατεβούμε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ε, όπως θέλει. Παρακαλώ. Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών. Και μια που προχωράτε προς το Προεδρείο σας. Καλώς ορίζω στην Νέα Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προσβλέπουμε πάρα πολύ στη συνεργασία μαζί σας τα επόμενα πέντε χρόνια και βέβαια να ευλογείτε πάντα αυτά που λέμε εμείς και να συμφωνείτε με τις απόψεις μας. So, so Λοιπόν, το μικρόφωνο και η θέση είναι δικιά σας κύριε Ρόιτε. Mm. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Για να δείξω στους συναδέλφους ότι μιλάω γερμανικά, θα αρχίσω στα γερμανικά και μην ανησυχείτε και θέλω να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος Γενικής Διεύθυνσης συνολικά αλλά και του Αντιπρόεδρου κυρίου Ταγιάννη και να σας συγχαρώ στο διορισμό στην Επιτροπή αυτή ως Πρόεδρο και βεβαίως και τους αντιπρόεδρους. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πάλι ενώπιόν σας και έχουμε την ευκαιρία να ξαναβλέπουμε πολλούς ε, γνωστούς ε, συναδέλφους, αλλά βλέπω και πολλά νέα πρόσωπα για μένα. Και χαίρομαι ήδη πάρα πολύ ε, και προσβλέπω στη συνεργασία μας το επόμενο διάστημα. Η Επιτροπή αυτή, θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα από την αρχή, ότι μπορεί να είναι εκείνη η Επιτροπή που, αν δούμε από στατιστικής απόψεως, κάνει την περισσότερη δουλειά ε, δίπλα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περίπου το 10% όλων των ε, διαδικασιών συναπόφασης στο παρελθόν ήταν εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών. Αυτό τι σημαίνει. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές και καινούρια μέλη, δεν διαλέξατε και την ευκολότερη Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Είναι όμως από τις πιο συναρπαστικές. Τα τελευταία χρόνια είχαμε μια πολύ καλή παράδοση ε, της συνεργασίας με εμπιστοσύνη και αυτό που έχω να σας προσφέρω και θέλω να σας προσφέρω να συνεχίσουμε υπό την έννοια αυτή τη συνεργασία μας και στο νέο κοινοβούλιο. Οι συνεργάτες μου και εγώ είμαστε στη διάθεσή σας για όλα τα θέματα Πολλοί από τους παλιούς συναδέλφους γνωρίζουν ότι είμαστε πάρα πολύ προσβάσιμοι. Αυτό σημαίνει ότι συμφωνούμε πάντα. αυτή είναι άλλωστε και η διαδικασία η δημοκρατική. Ε, υπάρχει και μια άλλη λοτριβή κάποια στιγμή για να προσπαθήσουμε να βρούμε τις καλύτερες προτάσεις. Να τα πω τώρα στα αγγλικά, γιατί αρκετά γερμανικά μίλησα. Um, Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας δώσω μία πρώτη εικόνα αυτών που φανταζόμαστε ότι θα εγγραφούν στην ημέρα της Επιτροπής σας τους επόμενους μήνες. Πρέπει να σας πω ότι είμαι σε ευαίσθητη θέση γιατί αυτή τη στιγμή γίνονται αλλαγές στην Επιτροπή και επομένως κατά αυτή την έννοια θα ήθελα να περιοριστώ ε, στην αναφορά συγκεκριμένων ε, υφισταμένων προγραμμάτων και όχι για μελλοντικές στρατηγικές. Όμως ε, είμαι ευτυχής γιατί μπορώ να μιλήσω για συγκεκριμένα ντοσιέ τα οποία αφορούν όμως το μέλλον των μεταφορών η Ευρωπαϊκή, που, που έχει εγκρίνει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να επικεντρωθώ σε αυτό. Εάν μου επιτρέπετε, Υπάρχουν ε, τρία πράγματα, τρία, τρεις λέξεις που στα αγγλικά αρχίζουν από C. Citizens, οι πολίτες, climate change, κλιματική αλλαγή και competitiveness, ανταγωνιστικότητα. Αυτά είναι τα τρία C που οδηγούν ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς μπορείτε να βρείτε και άλλα στοιχεία βέβαια, αλλά βάσει αυτών των τριών ε, αγγλικών C έχουμε προσπαθήσει, γύρω από αυτά τα τρία C, έχουμε υφάνει την πολιτική μεταφορών. προσπαθούμε να επικεντρώσουμε στην ανταγωνιστικότητα, γιατί οι ε, μεταφορές αποτελούν 7% του ΑΕΠ, 5% των συνολικών θέσεων απασχόλησης. Στο πρώτο C υπάρχουν τρία Ι. αγγλικά. Infrastructure, υποδομή, innovation, καινοτομία, internal market, εσωτερική αγορά. Και νομίζω ότι με αυτά που σας είπα έχουμε μια πρώτη ιδέα για το τι σημαίνει η ε, ε, πολιτική μεταφορών όσον αφορά την βιομηχανία, όσον αφορά την εξωτερική θεώρηση και την, τον εξωτερικό αντίκτυπο. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο C, climate change, κλιματική αλλαγή, πρέπει να ε, συνειδητοποιήσουμε ότι οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν ένα τέταρτο όλων των εκπομπών θερμοκηπίου. Και επομένως και όσον αφορά τις ε, ε, κλιματικές αλλαγές ε, έχουμε ασχοληθεί με πάρα πολλά επιμέρους θέματα, όχι όμως με τις μεταφορές. Από τη δεκαετία του 90 η συμβολή <clears throat> των μεταφορών στο φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει αυξηθεί πλέον του 1 τρίτου. Και με τις μελλοντικές ε, διεργασίες της ε, Κοπενχάγης οι κλιματικές αλλαγές ε, θα αποτελέσουν σημαντικό όχημα των μεταφορών. Και βεβαίως και εδώ μπορεί κανείς να βρει κάποιες υποκατηγορίες σε αυτό το θέμα. Τρίτο στοιχείο είναι βεβαίως ο πολίτης. Ο πολίτης λοιπόν ως ε, εργαζόμενος στον τομέα των μεταφορών, αλλά και ως χρήστης των μεταφορών. Άρα, κοινωνική διάσταση. Διάσταση όσον αφορά την ασφάλεια και όσον αφορά τις ασφαλείς μεταφορές. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία τα οποία διέπουν την πολιτική των μεταφορών. Και σε αυτές τις τρεις αρχικές παραμέτρους που έθεσα, ο Αντιπρόεδρος ε, Ταγιάννη έχει ε, δημοσιεύσει ανακοίνωση για, για το μέλλον της πολιτικής μεταφορών, όπου βεβαίως ε, θα ακολουθήσουν τις μελλοντικές τάσεις της κοινωνίας. Ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουμε περικοπές των ε, δημοσίων δαπανών, λιγότερες δεξιότητες, ε, μετανάστευση, εσωτερική κινητικότητα, περιβαλλοντικές προκλήσεις, που μόλις ανέφερα άλλωστε. Αλλά, επίσης, και την συνειδητοποίηση ότι το πετρέλαιο ή τουλάχιστον πετρέλαιο σε λογική τιμή αρχίζει να εκλείπει. Θα μας λείψει λοιπόν το πετρέλαιο ή πετρέλαιο σε λογική τιμή. Και αυτά όλα στα επόμενα ίσως όχι 5 χρόνια αλλά 10 με 20 χρόνια σίγουρα και αυτό θα σημάνει ριζική αλλαγή, ρήξη θα μπορούσα να πω, στο, στα υφιστάμενα συστήματα μεταφορών. Αυτά είναι τα στοιχεία προς σκέψη όσον αφορά τις μεταφορές. Η αστικοποίηση είναι επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Έχουμε αυξανόμενη ροή ε, προς τα αστικά κέντρα. Αυτό σημαίνει περισσότερη μόλυνση και περισσότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η παγκοσμιοποίηση επίσης ε, και παγκοσμιοποίηση όσον αφορά και την μεταφορά αγαθών και τη μετακίνηση εργαζομένων ε, και όσον αφορά την μηχανοκίνηση των μεταφορών γενικότερα. Και αυτά είναι στοιχεία προς σκέψη. Όλοι λοιπόν μέχρι ένα βαθμό εσείς σαν Κοινοβούλιο, εμείς σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν ορισμένα ριζικά ερωτήματα όσον αφορά την πολιτική μεταφορών για τα επόμενα χρόνια. Και το κύριο μήνυμά μου προς εσάς σήμερα είναι το εξής. Υπάρχει επιλογή. Επιλογή για όσους πολιτικούς ασχολούνται με τις μεταφορές και για αυτούς που γενικώ ασχολούνται με τις μεταφορές να καθορίσουν την μελλοντική ατζέντα ή να αφήσουν τους ανθρώπους της ενέργειας, ε, των τραπεζών ε, ή της οικονομίας ε, να καθορίσουν την ατζέντα των μεταφορών. Εγώ προτείνω να συνεργαστούμε τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε ο ομού ως ασχολούμενοι με τις μεταφορές να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις που είναι βεβαίως και πρόκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, όμως πρέπει να πω ότι πολλές από τις απαντήσεις θα πρέπει να εξευρεθούν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Άρα θα πρέπει να συνεργαστούμε και με αυτή τη λέξη την τρομερή που αρχίζει από S, subsidiarity, επικουρικότητα. On regional Επομένως, ναι, να σκεφτούμε ευρωπαϊκά, αλλά να ενεργήσουμε και τοπικά ή περιφερειακά. Επομένως, κατά αυτήν την έννοια θα ε, προωθήσουμε τις συζητήσεις μας τους επόμενους μήνες και χρόνια. Επί τη βάση αυτής ε, της ε, συζητήσεως σχετικά με το μέλλον της ε, πολιτικής μεταφορών, επί τη βάση του δικού σας feedback, των δικών σας συζητήσεων, των δικών σας εισρωών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διατυπώσουμε μια νέα λευκή βίβλο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών και θα ήθελα να σας δώσω μια γεύση των συγκλονιστικών πραγμάτων που μας περιμένουν ε, εν ώψη της προσπάθειας αντιμετώπισης των τριών C της πολιτικής μεταφορών. Θα, θα ολοκληρώσω σύντομα κύριε Πρόεδρε και μετά βεβαίως θα είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήματα κάθε είδους. Πολύ σύντομα θα ήθελα να ασχοληθώ με ορισμένους φακέλους που πιστεύω ότι ε, θα είναι θέματα που θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξή σας τους επόμενους μήνες. Πρώτα απ' όλα και η κυρία Γιάλα Σέντερ ήδη ε, ρώτησε σχετικά. Ενδεχομένως ε, θα υποβάλλουμε νομοθεσία όσον αφορά ε, την όσον αφορά τα ατυχήματα της πολιτικής αεροπορίας. Είχαμε αρκετά ατυχήματα τα τελευταία χρόνια. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ε, χώρος ανάπτυξης ρόλου της ΕΑΣΑ στον τομέα αυτό, αλλά βεβαίως αυτό προϋποθέτει συντονισμό ανάμεσα στις εθνικές υπηρεσίες διερεύνησης ατυχημάτων. Επίσης, και ο Αντιπρόεδρος Ταγιάννη ε, αναφέρθηκε σε αυτό την 8η Σεπτεμβρίου μετά από το σημαντικό ατύχημα, συνδρομικό ατύχημα στο Βιαρέτζο θα ε, ε, υπάρξει μια διάσκεψη για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και θα προσκληθείτε βεβαίως στην διάσκεψη αυτή. Εμείς θα προωθήσουμε ε, σχέδιο δράσης ε, για την αστική κινητικότητα, urban mobility, μέσα στο Σεπτέμβριο. Αυτό θα είναι ένα σχέδιο δράσης ε, το οποίο στην ουσία θα ασχολείται με αυτά τα τρία C και με το ένα μεγάλο S, την subsidiarity, την επικουρικότητα. Αυτή τη στιγμή εσείς εξετάζετε και την νομοθεσία ε, για την ασφάλεια, για τα δικαιώματα συγγνώμη, των επιβατών σε κάθε μορφή μεταφορών. Έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις στο Συμβούλιο και φαίνεται ότι χρειαζόμαστε την βοήθειά σας όσον αφορά τον ε, στόχο της προτινόμενης ε, νομοθεσίας. Περιμένουμε ότι η πρόταση για τις θαλάσσιες λεωφόρους θα προωθεί στο Συμβούλιο Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο για δεύτερη ανάγνωση. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2009 βέβαια. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ε, σημαντική πρόταση έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ε, πρόσβαση και στις συνδρομικές μεταφορές ε, εμπορευμάτων μέσω αυτών των ε, διαδρόμων ε, μεταφορών. Και πρέπει να σας πω ότι με μεγάλη προσοχή άκουσα ε, και την ε, συζήτησή σας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών και τη στήριξη που όλοι δώσατε στην κυρία Γένσεν ε, για τις διαπραγματεύσεις και ο κύριος Καραμίτσος είπε προηγουμένως ότι ε, δουλεύουμε ήδη πάνω στο θέμα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι θυμάμαι ότι εγώ εθελοντικά είχα ασχοληθεί με το θέμα αυτό πριν από 10 χρόνια και μάλιστα είχα πει ότι και στην προκείμενη περίπτωση η εθελοντική προσέγγιση ήταν η καλύτερη αλλά φαίνεται ότι 10 χρόνια μετά χρειαζόμαστε δεσμευτική ε, νομοθεσία. Όσον αφορά τις, ε, την εξωτερική πολιτική, όσον αφορά την ενδυνάμωση της συνεργασίας ε, στα θέματα μεταφορών ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αφρική. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, οδική ασφάλεια, ε, συνεργασία όσον αφορά τις ναυτικές ε, θαλάσσιες μεταφορές. Αυτά είναι ε, σημαντικά στοιχεία. Και βεβαίως, βεβαίως έχετε μπροστά σας και μία υποσχεθήσα πρόταση σχετικά με την χρηματοδότηση της ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύριο θα εγκρίνει απόφαση σχετικά με την επιμήκυνση της εντολής των συντονιστών των ΤΕΝΤΗ. Και επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια, δηλαδή ότι είμαστε όλοι ε, πραγματικά συντετριμένοι από τον ευνίδιο θάνατο του Καρλ Βαν ο οποίος συντόνιζε τα θέματα των μεταφορών. Ο Κάρλ ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε ασχοληθεί τόσο ενεργά με, την επιτρο... με, το... θέμα των μεταφορών, την πολιτική μεταφορών. Ήταν ο πρώτος ο οποίος παρήγε ε, ε, λευκή ε, βίβλο. ήταν αυτός ο οποίος στην ουσία δημιούργησε ε, την DG Transport, την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και την έκανε, τη μεταμόρφωσε σε μια Γενική Διεύθυνση η οποία ασχολείται πραγματικά με την ουσιαστική πολιτική των μεταφορών. Ήταν καλός φίλος όλα αυτά τα χρόνια και ε, πραγματικά ε, πρέπει να σας πω ότι είμαστε όλοι εξαιρετικά λυπημένοι. Βεβαίως θα αντικατασταθεί ο, ο κύριος Βαν ε, ο, ο, ο Βαν καθώς επίσης και ο κύριος Μπάλας. Υπάρχουν ε, και άλλα τεχνικά μέτρα τα οποία θα έρθουν προς εσάς. Ε, η αναθεώρηση σχετικά με τον οδικό εξοπλισμό, τον θαλάσσιο εξοπλισμό και πολλά στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά σχετικά με τον ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο δεν πρόκειται για τεχνική πρόταση, είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρόταση η οποία αφορά τον τρόπο λειτουργίας των θαλασσίων λεωφόρων. Το να πάει κανείς, ας πούμε, από την Κοπενχάγη στον ε, Πειραιά ε, δεν μπορεί να γίνει μονάχα με φορτηγά. Θα πρέπει να μπορεί να γίνεται ε, με απλό τρόπο και διαθαλάσσεις στα πλαίσια του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου. Πρέπει να σας πω ότι η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών πάντα θεωρούσε ότι η Επιτροπή σας είναι σημαντικό στήριγμα και το απέδειξε επανειλημμένα. Μπορώ να αναφέρω εδώ το ζήτημα της χρηματοδότησης των διευρωπαϊκών δικτύων. Μπορώ να αναφέρω εδώ και ένα πιο αντιφατικό, ε, αφιλεγόμενο μάλλον ζήτημα, ε, που είναι οι ώρες εργασίας των εργαζόμενων στις οδικές μεταφορές. Πολλά έχουμε και μπροστά μας, πολλά δύσκολα μας περιμένουν και πραγματικά περιμένω από την Επιτροπή σας να συνεχίσει την συνεργασία μαζί μας, με τη Γενική Διεύθυνση μαζί μας, με τον ευφυή e e και ορθό τρόπο με τον οποίο συνεργαστήκαμε τα τελευταία χρόνια. Έχετε κάνει πάρα πολλή δουλειά, πολύ σημαντική δουλειά και εδώ σας ε, ε, δίνω και ένα βιβλίο το οποίο αναφέρει τι έχει κάνει και η Επιτροπή το τελευταίο, καιρό. Και θα είμαστε πάντα ο ένας δίπλα στον άλλον, ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε τόσο νωρίς, τόσο γρήγορα στην Επιτροπή μας. Θα συμφωνήσουν οι συνάδελφοι ότι προσβλέπουμε μονησία στη συνεργασία με εσά και το προσωπικό της υπηρεσίας σας. Ο κοινός στόχος είναι αναβάθμιση των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ο εντοπισμός των ευρύτερων ευθυνών που έχουμε για τις πόλεις και για το ε, κλίμα, για τις κλιματικές αλλαγές. Έχουμε διάφορους ομιλητές. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω την ε, λέξη που αρχίζει από D, ε, discipline, πειθαρχία. Θα προσπαθήσω να επιβάλλω κάποια πειθαρχία ως προς το χρόνο αγόρευσης. Παρακαλώ να είστε ως το δυνατόν πιο σύντομοι και περιεκτικοί γίνεται. Έτσι θα μας βοηθήσετε. Ας αρχίσουμε με τους συντονιστές και μετά θα περάσουμε στα μέλη της Επιτροπής. Έχετε κατά νου το χρόνο, τον περιορισμένο χρόνο που έχουμε, γιατί θέλουμε όλοι να περάσουμε ένα μήνυμα στον Γενικό Διευθυντή και θέλουμε πρέπει να το αφήσουμε και χρόνο απαντήσεις στη συνέχεια. Ο κύριος Γκρόσε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την παράδοση να ε, ξεκινούν οι συντονιστέ, αλλά θα είμαι για να μιλήσουν και οι συνάδελφοι, όχι μόνο οι συντονιστέ. Ευχαριστώ. Δεν είναι εύκολο το έργο σα Στην αρχή μια κοινοβουλευτική περίοδου να έρχεστε έτσι γρήγορα γρήγορα μα δίνετε μια μεγάλη επισκόπηση. Ούτε θέλω να υπογραμμίσω όλα όσα είπατε. Γνωριζόμαστε και από το παρελθόν, ξέρουμε τις προκλήσεις, κλίμα, ενέργεια, κινητικότητα, ε, ασφάλεια κτλ. Ε, τρία σημεία θέλω να τονίσω. Πρώτον, όλοι όσοι είμαστε σε επαφή με τις μεταφορές, επιτόπου δηλαδή, βλέπουμε ότι σήμερα, αλλά και πριν από μερικούς μήνες, βλέπαμε να αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα της λεγόμενης οικονομικής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει πρωτοβουλία εδώ σε αυτό το θέμα στους διάφορους τομείς για να δώσει οθήσει προβληματισμού δυνατότητες, γιατί υπάρχουν και προσδοκίες προς εμάς δεν λέω ότι περιμένουν λιγότερους κανόνες, αλλά κάποια κατανόηση για την κατάσταση που ζουν. Το ένα αυτό. Το δεύτερο αφορά ένα άλλο C που είναι communication, η επικοινωνία. Νομίζω ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά σε αυτό το τομέα και δείξαμε και μεγάλη πειθαρχία ε, στην προεκλογική εκστρατεία και διαπιστώσαμε ότι προς τα έξω ε, δεν φτάνει και το μήνυμα στο βαθμό που θα επιθυμούσαμε. Παρόλο που έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ σκληρά με αυτά τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν μπορούμε από κοινού, Βούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να διαμορφώσουμε την κοινωνία μας έτσι, ε, ώστε να την καταλαβαίνουν όλοι και όχι τα μέλη εδώ της Επιτροπής ή οι ειδικοί που ζουν και ε, δουλεύουν. Και ε, το τελευταίο, το αγαπημένο μου θέμα που είναι να μαλώνω το Συμβούλιο. Ε, είναι πολύ καλές ιδέες αυτές που εμεί αποφασίζουμε και τη συναποφασίζει και το Συμβούλιο, τονίζω, ε, απέχουν πολύ από τα όσα συμβαίνουν στα κράτη-μέλη, γιατί και εκεί χωλαίνει η κατανόηση των πολιτών. Δηλαδή, όταν λέμε, μα κοιτάξτε, αποφασίσαμε το α ή το β, και ε, οι πρώτοι ψάχνουν ε, εξαιρέσεις, οι δεύτεροι δεν το εφαρμόζουν καθόλου και οι τρίτοι το εφαρμόζουν με τρόπο ε, πολύ περίπλοκο και ερχόμαστε και μετανιώνουμε πικρά σχεδόν που ανοίξαμε καν το θέμα αυτό. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσαμε να το ξαναδούμε. Κάποια πράγματα που αποφασίσαμε στο παρελθόν. Μήπω χρειάζεται απλούστευση, μήπω χρειάζεται βελτίωση, χωρί να ανοίξουμε τώρα τι πόρτε για όλα τα θέματα ήθελα να το τονίσω γιατί ε, τα άλλα τα ενδιαφέροντα τα είπατε εσείς, ίσως είναι κάτι παραπάνω αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κύριος Λάιχτφριντ. Ευχαριστώ. Κύριε Γενικέ, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε τόσο νωρί στην Επιτροπή μας και μας είπατε τόσο ενδιαφέροντα πράγματα. Και εγώ να επικεντρωθώ σε τρία ζητήματα και να περιοριστώ. Το πρώτο πακέτο ερωτήσεων αφορά την ασφάλεια των αερομεταφορών η κατάσταση είναι ικτρή. Πραγματικά, ο κόσμος που πετάει ταλαιπωρείται. Το ψάχνουμε στις κρέμες του, τι είναι αυτά τα δολοφονικά όπλα που κυκλοφορεί, τη ε, κρέμα ξυρίσματος και τα παίρνουμε και με επιτυχία και μετά πέφτουν αεροπλάνα. Ε, ξέρω εγώ μήπως ε, αρμενίζουμε στραβά. Πώς θα συνεχίσει η ιστορία αυτή με τα υγρά. Και μετά τι συγκεκριμένα θα κάνετε έτσι ώστε στην Ευρώπη να είναι πιο ασφαλής οι αερομεταφορές, η κυκλοφορία. Θα υπάρξει ε, κάποιος έλεγχος και στις ευρωπαϊκές εταιρείες γιατί οι επιβάτες πολύ ταλαιπωρούνται. Και είναι πολύ μεγάλη αβεβαιότητα και ανασφάλεια και θα πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Ε, δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σχεδιάζει συγκεκριμένα για να γίνει πιο οικολογική ε, η συγκοινωνία γενικά. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι έχουμε προβλήματα με την οικονομική κρίση. Αλλά σιγά σιγά δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθεί προγράμματα για πιο εντατική ε, κυκλοφορία των φορτηγών. Αυτό είναι η απάντηση στην οικονομική κρίση, να ενταθεί η κυκλοφορία των φορτηγών στους αυτοκινητοδρόμους. Μήπως θα πρέπει να πάμε σε άλλα οικολογικά συστήματα μεταφοράς. Και εδώ πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, ε, σε σχέση και με τη Σουηδική Προεδρία κυκλοφορούν διάφορες φήμες ότι λέει θα προσπαθήσουν να κάνουν νέες ρυθμίσεις. Πριν από δυόμιση χρόνια εμείς αποφασίσαμε ήδη κάτι που έχει νόημα και με συναδέλφους από άλλες πολιτικές ομάδες το έχουμε συζητήσει. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενδιαφέρεται να ξανανοίξει αυτό το θέμα. Και ένα τρίτο έχετε κυρίως ή αποκλειστικά προγράμματα μεταφορών θήξη και μιλήσετε μόνο για τις μεταφορές. Η Επιτροπή μας ασχολείται και με τον τουρισμό. Εκεί τι έχουμε. Και κυρίως τι γίνεται η ιστορία αυτή με τις βινιέτες στα σήματα κυκλοφορίας στη Σλοβενία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λάιχφριτ. Ο κύριος Στέρξ από τους Φιλελευθέρους για τρία λεπτά. Συντονιστές τρία λεπτά και λυπή δύο, έτσι για να έχετε μια ιδέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ρόιτερ, που ήρθατε και τόσο γρήγορα μετά τις εκλογές ε, στη νέα Επιτροπή Μεταφορών για να έχουμε και το γενικό πλαίσιο. Ήδη από την αρχή είπατε ότι είναι δύσκολη η καιρή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ενδεχομένω αλλάζει και επίτροπος. Ε, και ο σημερινό επίτροπο ε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ίσω θα επιβεβαιωθεί τι θα έρθει άλλο. Οπότε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό είναι δύσκολο. Ένα σημείο που δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο του, χρόνου θα χρειαστεί νέα ε, λευκή βίβλος αρχέ του χρόνου και όποιο επίτροπος και να είναι παλιό ή καινούριο, θα πρέπει να προετοιμάσει αυτή τη λευκή βίβλο. Και τώρα έχουμε και ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής για τι κατευθυντήριε γραμμέ, ε, κάπου θα πρέπει να προσανατολιστούμε, όποιο και να είναι ο επίτροπο, για τι κατευθυντήριε γραμμέ για την πολιτική μεταφορών. Έτσι, να χαραχτούν από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Υποθέτω ότι αφορά και το Συμβούλιο αυτό. Η φιλοδοξία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη, ελπίζω. Και οπωσδήποτε από την Επιτροπή θα πρέπει να έχουμε προσέγγιση όσο γίνεται πιο ευρωπαϊκή. Τουλάχιστον αυτό εμείς περιμένουμε από την ε, Κομισιόν. Τι σημαίνει αυτό. Γενικά, αηφορία, έτσι κι αλλιώς, ε, ένας βιώσιμος κλάδος μεταφορών και από πλευράς οικονομικής και κοινωνικής και οικολογικής, γιατί δεν έχει νόημα εκεί να διαταράξουμε τις ισορροπίες ή να τις βάλουμε λάθος, ε, πραγματικά προσβλέπω με μεγάλο ενδιαφέρον ε, τι θα κάνετε. Στην ανακοίνωση αναφέρονται μερικά θέματα αρκετά ενδιαφέροντα. Ε, το επόμενο διάστημα σίγουρα θα προχωρήσουμε έτσι κι αλλιώς. Και αυτό που θέλουμε να τονίσουμε εμείς είναι η διάνοιξη των αγορών. Δηλαδή, να δούμε την αγορά ευρωπαϊκή για όλα τα μέσα μεταφορών και να πέσουν τα εμπόδια που δυστυχώς είναι ακόμα μεγάλη. Μιλήσατε για τον Κάλβαν Μιρθ και σας ευχαριστώ γιατί ήταν συμπατριώτης μου. Ξεκίνησε αυτή τη δουλειά, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά και όλα αυτά τα χρόνια ότι κάθε φορά που θέλουμε να φτάσουμε σε συμφωνία, Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μαζί απέναντι στο Συμβούλιο. Κάθε φορά τους βγάζουμε με το τσιγκέλι μια συμφωνία και φτύνουμε αίμα. Τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια λοιπόν. Και στην Επιτροπή Μεταφορών ελπίζω να υπάρξει μεγάλη πλειοψηφία προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Ευχαριστώ, Dirk. Από του Πρασίνους, ο κύριος Κράμε. Ευχαριστώ. Και τώρα, κατάλαβα γιατί τα είπατε ε, ε, ε, αγγλικά, γιατί τα τρία C είναι πιο ωραία από το P και V που είναι τα αρχικά στα γερμανικά και δεν σας βγαίνανε. Λοιπόν, για την προστασία του κλίματος είπατε ότι το 1 τρίτο ε, των εκπομπών διοξιδίου βγαίνουν ε, από τις μεταφορές και αύξηση 35% έχουμε από τη δεκαετία του 90. Αυτό έρχεται να οξυνθεί, αν δείτε ότι σε όλους τους άλλους τομείς έχουν μειωθεί κατά 10% οι εκπομπές. Δηλαδή ό,τι εξοικονομούμε στη θερμομόνωση, στη βιομηχανία με δισεκατομμύρια επενδύσεων, τα τρώει όλα ε, το σύστημα των μεταφορών. Λοιπόν, αν δεν αλλάξουμε τις μεταφορές, δεν πρόκειται να προστατεύσουμε το κλίμα και να ε, αλλάξουμε την κλιματική αλλαγή εμείς. Τα είπατε ξεκάθαρα και σας ευχαριστώ. Επίσης είπατε ότι μας τελειώνει το πετρέλαιο αν έχουμε 450 αυτοκίνητα σε χίλιους ε, κατοίκους, οι Ρώσοι είναι 170 αυτοκίνητα και οι Κινέζοι 15 στους χίλιους κατοίκους. Αν φτάσουν αυτοί στα 450, δεν θα μας τελειώσει το πετρέλαιο, θα σωθεί και το τσάλι και ό,τι άλλο θέλετε. Δεν θα έχουμε καμία πηγή ενέργειας. Αν τα βλέπουμε αυτά παγκόσμια, ε, πρέπει να αλλάξουμε λαγική και συμπεριφορά. Α, για την πόλη τώρα. Εκείνο όλη η εκπομπή κατά 70% πάλι προκαλούνται από τις κοινωνίες, τις αστικές μεταφορές και εκεί κάπως θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Ξέρω ότι υπάρχουν αντιστάσεις. Ένας μοχλός που μπορούμε να ε, επέμβουμε παρά την επικουρικότητα είναι το χρήμα. Και εδώ στο Κοινοβούλιο αποφασίσαμε στο μέλλον τουλάχιστον 40% των επενδύσεων στις μεταφορές να πάνε στο σιδηρόδρομο. 60% ε, σήμερα πηγαίνουν στο αυτοκινητόδρομο και 20% μόνο στο σιδηρόδρομο. Θα πρέπει να συμφωνήσει το Συμβούλιο και να τα υλοποιεί. Εσείς πώς προτίθεστε αυτή την απόφαση του Κοινοβουλίου να την κάνετε και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τελευταίο. Είναι πολύ φτηνές οι μεταφορές στην Ευρώπη. <coughs> και κάνουμε και πολλές βλακίες. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξάγει 5 εκατομμύρια ε, τόνους ε, ε, χειρίου κρέατος και εισάγει το ίδιο ποσό. Εδώ χρειάζεται φυΐα, όχι μεταφορές. Η Ευρώπη εξάγει κοτόπουλο στην Αφρική και είναι πιο φτηνό εκεί το κοτόπουλο, το ευρωπαϊκό, από ότι το αφρικανικό ντόπιο. Αυτό είναι τρελό και από πλευρά αναπτυξιακή πολιτική αλλά και από πλευρά μεταφορών. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και τέλο, όταν παίρνω το τρένο από το Βερολίνο στι Βρυξέλλε, παίρνω 19% ΦΠΑ και αν πάρω αεροπλάνο μηδέν, παρόλο που είναι τριπλάσια επικινδυνότητα των εκπομπών. Πού είναι ο υγιή ανταγωνισμό competition που είπατε. Είναι fair competition, όχι εστρέβλωση του ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, θα τελειώσουμε τον πρώτο γύρο. Θα ζητήσουμε απαντήσει από τον κύριο Ρόιτερ, ο κύριος Βαντάλιν προ το παρόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ρόιτερ που ήρθατε τόσο γρήγορα στην Επιτροπή μας και επίσης ευχαριστώ που μιλήσατε και για το τραγικό θάνατο του Καρλ Φανμίρτ στη δεκαετία του 80 ε, τον είχα ζήσει εγώ εδώ συνεργάτης και είδα πόσο ενθουσιώδης ήταν για τις μεταφορές στην Ευρώπη και πραγματικά μας λείπει πολύ. Τρία θέματα. Πρώτον, οι υποδομές. Ζούμε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης και υποχώρησης και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα προγράμματα συγχρηματοδότηση στα δύο ευρωπαϊκά δίκτυα. Δεν μπορούν να επιταχυνθούν οι διαδικασίε για να βοηθήσουμε και την οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη και την απασχόληση. Και θα ήθελα να παρακαλέσω να κοιτάξετε πάρα πολύ καλά αν υπάρχουν εκεί δυνατότητε χρηματοδότηση επιταχυμένη. Ε, ιδιαίτερα για την εσωτερική ναυσιπλοεία, για κάποιες προκαταβολές που δυστυχώς ε, πληρώνουν την ύφη στα δύο ευρωπαϊκά ε, προγράμματα. Δεύτερον, Κάτι που δεν άκουσα στην παρουσίασή σας είναι η υλοποίηση της νομοθεσίας. Ε, σκοπός δεν είναι να βγάζουμε κανόνες, αλλά να κοιτάμε πώς υλοποιούνται και με σωστό τρόπο. Παντού. Δεν είναι μόνο οι οδικές μεταφορές. Και το, οι μετακινήσεις το καλοκαίρι. Ας πούμε στην Ιταλία τους βάζουν τεράστια πρόστιμα σε συμπολίτες μας ε, Ολλανδούς για παραβιάσεις ε, μικρές του κώδικα δικής ε, κυκλοφορίας. Τι γίνεται με το στρέβλος ανταγωνισμού, τι γίνεται με την υλοποίηση των όσων αποφασίζουμε κτλ. Και τέλος επικουρικότητα. Η δική μου πολιτική ομάδα ενδιαφέρεται πάρα πολύ με αυτό το θέμα και ρωτώ θα πρέπει ε, να μελετάμε τον αντίκτυπο κάποιων αποφάσεων ευρωπαϊκών σε συγκεκριμένες περιοχές. Ας πούμε, ε, στα νησιά της Σκοτίας λέει ε, κάποιος ακτοπλός ότι θέλει να βάλει δρομολόγιο και την Κυριακή. Οι κάτοικοι λένε δεν μας χρειάζεται. Λοιπόν, ποιος έχει δίκιο. Αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα και ξέρουν τι γίνεται και εκείνη η επικουρικότητα ή θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να επιβάλλει τον κανόνα του οκτοπλώ ε, εν ονόματι του ε, ανταγωνισμού. Αυτά τα θέματα είναι σημαντικά και χρειάζονται ειδική προσοχή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Βαντάλεν. Ο κύριος Ρόιτερ, θέλετε να αρχίσετε να απαντάτε την πρώτη δέσμη ερωτήσεων και μετά θα ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις και παρατηρήσεις από τα λοιπά μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο γιατί ανέφεραν σημεία που έπρεπε να είχα αναφέρει ο ίδιος ε, νωρίτερα. Ο κύριος Γκρός, όλος ιδιαίτερος σαφώς, ε, περιέγραψε την τωρινή κατάσταση, δηλαδή την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε σαφέστατα και στον τομέα των μεταφορών, ε, κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Είναι σαφής η κρίση και έχουμε ήδη προτείνει μια σειρά μέτρων ε, για τη μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων. Ακόμη ε, στα πλαίσια του κανόνα use it or lose it, ε, δηλαδή να χάνουν τα κονδύλια αν δεν απορροφούνται, κυρίως στην πολιτική αεροπορία. Το είπε και ο κύριος Βαντάλεξ εξάλλου. Για την εσωτερική ναυσιπλοεία που πλήττεται βαρέως ε, διότι όπως περιγράψατε και ε, πλήττονται όλοι οι τομείς ουσιαστικά. Το βασικό μήνυμα που εμείς περνάμε είναι να μην επαναχωρήσουμε, να μην καρκινοβατήσουμε πίσω τον προστατευτισμό. Έχουμε μια κατάσταση στην οποία καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε, μας κάνουμε ότι μπορούμε, αλλά μην επιστρέψουμε σε προστατευτικά μέτρα που ε, εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τώρα, ως προς την υλοποίηση, κάτι που έθιξαν διάφοροι συνάδελφοι, ναι, απαντώ, εν μελλοντικών εργασιών της Δέλτα τρέν είναι σαφώς σαφές ότι περισσότερο από το παρελθόν πρέπει να ρίξουμε το βάρος στην υλοποίηση της νομοθεσίας, στη μεταφορά μάλλον της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην νομοθεσία των κρατών μελών. Θα σας ενημερώσουμε για τις διαδικασίες επί παραβάση Προς το παρόν εξετάζουμε το όλο θέμα της υλοποίησης του σιδηροδρομικού πακέτου. Κάνουμε τακτικές εκθέσεις ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας, τις οποίες σας υποβάλλουμε. Αλλά όντως πρέπει να ε, δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό στην επόμενη περίοδο. Να μην έχουμε περισσότερες νομοθετικές πράξεις. Καλύτερα είναι να μεριμνήσουμε η υφιστάμενη νομοθεσία να εφαρμόζεται καλύτερα. Δεύτερον, ε, κύριε Γκρός, θίξατε ε, ένα επίσης ε, σημαντικό ζήτημα, αυτό της ε, απλούστευσης. Ε, υπολείπεται δουλειά. Πρέπει να συνεχίσουμε να εξετάζουμε την νομοθεσία, είτε μιλάμε για ενοποίηση του πρώτου συνδρομικού πακέτου, είτε μιλάμε για άλλα στοιχεία. να δούμε πού μπορούμε να επιφέρουμε απλούστευση στην νομοθεσία. Εργαζόμαστε από αυτού ήδη. επικοινωνία, communication, το τρίτο C και μάλλον είναι και το πιο σημαντικό. Το τέταρτο C μάλλον, που είναι το πιο σημαντικό. Ό,τι κάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, που είναι θετικό και το εκτιμούν οι πολίτες, δεν ε, αντιμετωπίζεται σαν, ε, ως ευρωπαϊκό, δεν θεωρείται ευρωπαϊκό. Ό,τι είναι επαχθές και δυσχερές, αυτό αντίθετα αναγνωρίζεται ως ευρωπαϊκό. Ε, η έλεγχη, ατελείωτη έλεγχη παραδείγματος χάρη. Πρέπει να, το, να δούμε το θέμα της επικοινωνίας. Για τα υγρά τώρα, κύριε Λάιχφριντ, στα αεροδρόμια. Πώς να το θέσω. Έχουμε αναλάβει ισχυρή δέσμευση. Ο αντιπρόεδρος Μπαρό ο Αντιπρόεδρος Ταγιάννη έχουν αναλάβει σαφώς τη δέσμευση να ε, κάνουν μια εισήγηση για τα υγρά. Ταυτόχρονα όμως ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε και την απαιτούμενη τεχνολογία για να τα φέρουμε, για να τα υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Ο Αντιπρόεδρος Ταγιάννη τις προσεχείς εβδομάδες και τις προσεχείς μήνες ε, θα ασχοληθεί με το θέμα και θα κάνει ανακοινώσει. Συμφωνώ πλήρως με τον Αντιπρόεδρο για αυτό το θέμα. Έχουμε μία δέσμευση να καταργήσουμε τον κανόνα για τον έλεγχο των υγρών, το screening. Ε, ταυτόχρονα όμως πρέπει να βρούμε τρόπους για να το κάνουμε αυτό χωρίς να έχουμε 27 διαφορετικούς κανόνες στα 27 κράτη-μέλη που θα είναι ακόμη επαχθέστερη για τους ε, πολίτες. Πρέπει να συνεργαστούμε δηλαδή για να βρούμε μια διέξοδο. Ο Αντιπρόεδρος ε, Ταγιάννη, υπό ειδικής προεδρία ε, δεν αναμένεται να κάνει πρόταση για, τις ε, μεγάλες, ε, για τα μεγάλα φορτηγά. Και υπάρχουν και άλλα στοιχεία της οδηγίας. Εξάλλου έγινε και ακρόαση, θα το θυμάστε. Νόμιζα θα ξεφύγω όταν μιλούσατε για τον τουρισμό. Mm λέγοντας ότι δεν είναι δική μας δουλειά, της δικής μας γενικής διεύθυνσης. Αλλά όταν αναφερθήκατε στη βινιέτα της Σλοβενίας, ε, σε ένα ορισμένο βαθμό θα έλεγα ότι είναι μεικτή αρμοδιότητα. Αλλά θα εξετάζουμε προσεκτικά το θέμα και σημειώνουμε αυτό που μας είπατε. Κύριε Στέρξ, το άνοιγμα της αγοράς σαφώς είναι ένα, ε, μία από τις ε, ε, κινητήρες δυνάμεις της ολοκληρωμένης πολιτικής μεταφορών ναι, και γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό που το θίξατε το θέμα. Κύριε Κάρμα, το γενικότερο ερώτημα, το γενικότερο θέμα της ε, πολιτικής ε, μεταφορών. Κοιτάξτε, τους ε, επόμενους μήνες, και ελπίζω δεν θα κρατήσει πολύ η διαδικασία, θα γίνει μεγάλη συζήτηση για την Ευρωβινιέτα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς πρέπει να χειριζόμαστε τα θέματα μεταφορών. Ο κύριος Αλκαντρόη αγωνίζεται σκληρά ε, για να υπεραμεινθεί τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Τώρα πρέπει να δούμε ε, πού θα καταλήξει τελικά αυτή η συζήτηση για την Ευρωβινιέτα. Κύριε Βαντάλεν, για την κινητοποίηση των κονδυλίων για την επίσπευση της ανάπτυξης υποδομής. Ναι, ε, ήδη με, στο σχέδιο ανάκαμψης οικονομίας με τα 500 εκατομμύρια ήδη έχουμε επιληφθεί του ζητήματος. σαφώς Ο λόγος ετοιμάτων προ τα κονδύλια είναι ένα προς τέσσερα και δεν έχουμε επαρκή κονδύλια. Ευχαριστούμε κύριε Ρόιτερ. Εννιά μέλη της Επιτροπής θέλουν να μιλήσουν. Θα διαβάσω τα ονόματα. Mr. Mr. Grandes Mr. Mr. Θα κλείσω το κατάλογο των ομιλητών και παρακαλώ, παρακαλώ να είστε όσο το δυνατόν συντομότεροι γίνεται. 1,5 λεπτό, το όριο, 2 λεπτά. Όταν αρχίζω να ε, ε, κουνάω το σφυράκι μου, ε, παρακαλώ να σταματήσετε αυτό πειθαρχηθείτε και θα σας είμαι ευγνώμονος, Πρόεδρος. Ο κύριος Κόκ. Κοκ, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ρούτε, τα εξή τρία και θα παρακαλούσα να εμβαθύνετε. Πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια. Δεύτερον, ε, μέτρα και σταθμά και βάρος των ε, φορτηγών και το κταίο, η τεχνική ε, μελέτη, παρακολούθηση και τα λεγόμενα ευφύ αυτοκίνητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κόχο. Ο κύριος Ελχαντράουι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι λίγο πιο μακροσκελής από τον κύριο Κόχο. Ευχαριστώ τον κύριο Ρούτε για την παρουσίασή του. Περιγράψατε κυρίως αυτά που γράφει η ανακοίνωση. Ωραία, τις μεγάλες προκλήσεις και ό,τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τη Λευκή Βίβλο. Θα πρέπει η Λευκή Βίβλος να είναι όσο γίνεται πιο συγκεκριμένη και κατά προτίμηση να συνδέεται και με ένα συγκεκριμένο χρόνο διάγραμμα για να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε και προς τα πού και πότε. Ε, υπό την έννοια αυτή μου τράβηξε την προσοχή κάτι ακόμα. Στην αξιολόγηση τονίζεται ότι είναι πρόβλημα, λέει, οι αηφόρες μεταφορές, ότι δεν φτάσαμε τους στόχους μας εκεί και παραπέμπεται στην Ευρωβινιέτα. Κοραστήκαμε πάρα πολύ και μαζί έχουμε και την ίδια θέση πάνω κάτω για να έχουμε φιλόδοξο πρόγραμμα εκεί και φιλόδοξη νομοθεσία. Τώρα φοβούμαι ότι στο Συμβούλιο έχει οδηγηθεί σε εμπλοκή. Δεν έχω την ε, αίσθηση ότι έχει κατενθουσιαστεί το Συμβούλιο να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Ερωτώ, μπορούμε να σκεφτούμε έναν τρόπο μαζί να κινήσουμε το Συμβούλιο να κάνει πρόοδος. Ε, εσωτερική του εξωτερικού κόστους μπορεί να είναι αυτό το στοιχείο κλειδί για να φτάσουμε στην αεφορία. Και μια συμπληρωματική ερώτηση που συνδέεται με το προηγούμενο. Στο περιθώριο της συζήτησης λέτε ότι θα έρθει με πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους κανόνες που θα τους ειδικού φόρους κατανάλωσης. Και εκεί θα έχετε συμπεριλάβει και το κόστος του διεξουδίου του άνθρακα των εκπομπών. Πώς έχει προχωρήσει αυτό. Και τέλος, μια μικρή επιφύλαξη που έχω για τη χρηματοδότηση της φύλαξης των αεροδρομίων και το πρόγραμμα δράσης. Το θέμα είναι, στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα που η ίδια έχει βάλει στον εαυτό της. Είναι δύο προτάσεις που ήρθαν ένα εξάμεινο κατόπιν εορτή. Στο μέλλον θα τα αλλάξετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Περίπου θα σας έπεφτε το σφυράκι κύριε κυρία Κύριε κυρία λοιπόν, έχω σημειώσει πολλά ερωτήματα σύντομα όμως. Πρώτον, το ζήτημα των επικινδύνων θέσεων στα αυτοκίνητα για βρέφη και μικρά παιδιά. Μας είπατε μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα φέρετε τη μελέτη. Πότε επιτέλου, Δεύτερον, gigaliners. Για μένα αυτό είναι προβληματικό. Δεν υπάρχει βουλευτής ε, που να είχε ορκιστεί, ας πούμε, πάνω κάτω. Μόλις πρώτο ήρθε έγινε μια παρουσίαση ε, που ήταν διαφήμιση του προγράμματος αυτού, αλλά υπάρχει και κοινωνικό κόστος για τα κράτη-μέλη, ε, για τα έργα. Και μη μας παρουσιάζουν αυτό το θέμα των gigaliners ως σούπερ επιτυχία. Θέλω να μου απαντήσετε σαφώς αυτό. Τρίτον, τα δικαιώματα των επιβατών στις αερομεταφορές. Ε, έγινε μια συζήτηση που ξεκίνησε για την άρνηση επιβίβασης, denied boarding Έχω την εντύπωση ότι όλο και περισσότεροι επιβάτες βγαίνουν και λένε ότι δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους και δεν είναι έτσι φτιαγμένα ώστε να μπορούν να τα επικαλούνται. Τρίτον, η κόπωση των ε, κυβερνητών. Έγινε μια μελέτη για τους χρόνους ανάπαυσης και οδήγησης και ό,τι αφορά την κόπωση και τις συνέπειες τους φαίνεται δεν έχει ετοιμαστεί η μελέτη. Θα πρέπει να τη συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή μας γιατί τη τελευταία θητεία κάναμε μια πολύ εντατική συζήτηση ε, στη συνέχεια ε, σε σχέση με τον αέρα που κυκλοφορεί στο εσωτερικό της ατράκτου. Πρέπει να λυθεί το θέμα. Είναι πολύ ανετικές ε, οι εμπειρίες. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς θα εφαρμόσετε τους ελέγχους στα φορτηγά. Τα κράτη-μέλη είναι τόσο αμελείς στους ελέγχους που επιδεινώνεται όλο και περισσότερο η ασφάλεια στους δρόμους. Ε, Ξέρετε τι με, με εκπλήσετε, τι γλιτώνετε κάθε φορά για κλάσματα δευτερολέπτου. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο του για την ε, άμεση έλευσή του και την παρουσίαση για την πληροφόρηση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και να επιμείνω στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Τι έγινε, χάθηκαν ε, κάποιες ρυθμίσεις για τις παραβάσεις και τι γίνεται εκεί, τι γίνεται και με την αξιολόγηση των στόχων ε, του 2010 και το νέο ε, πλάνο, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Γαλιλαίος. Ακούμε διάφορα πράγματα για διάφορα κέντρα. Στη συμφωνία είχαμε αποφασίσει για τρία. Μπορείτε να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό. Σας ευχαριστώ επίσης για το φόρο τιμής που αποτίσατε στον κύριο Κάλβαν Μίρτ και συμφωνώ απολύτως. Αύριο θα αντικατασταθούν δύο συντονιστές θα αλλάξει και ο κύριος Δαβινιών, ο οποίος είχε μια πολύ ατυχή εμφάνιση εδώ. Για την Αφρική, τι γίνεται με τη Σομαλία στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Τώρα ασχολούνται άλλες γενικές διευθύνσεις, αλληλεία, ξέρω εγώ και τα αλλά είναι και θέμα ασφάλειας στην αυσιπλοεία και στις μεταφορές. Η πειρατεία. Για τη χρηματοδότηση θα με ενδιαφέρει πολύ ε, να μάθω τι λέει η Γενική σας Διεύθυνση για τη Γενική Συζήτηση για το μέλλον, για τα ευρωπαϊκά δίκτυα αεροπορία, μιλάμε για την ασφάλεια, αλλά και για την υγεία και για την άνεση. Περίπου ο κόσμος ε, στηβάζεται και ε, η μεταφορά δεν είναι αξιοπρεπή σε πολλές περιπτώσεις. Επίσης η υλοποίηση, καλές οι ρυθμίσεις και τα μέτρα, αλλά η υλοποίηση θα πρέπει να είναι δεύτερη ευκαιρία για την ε, επικοινωνία να μην εφαρμόζουμε 27 διαφορετικά πράγματα, αλλά αυτό που αποφασίζεται να εφαρμόζεται και ενιαία. Ευχαριστώ πολύ. Τελειοποιήσατε την τέχνη εσείς. Ε, η κυρία Φώστερ, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον προσκεκλημένο μας που ήρθε σε τόσο πρώιμο στάδιο σε συνεδρίες Επιτροπής μας. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Το πρώτο ήταν για τα υγρά στα αεροπλάνα. Νομίζω ότι πολύ θα δυσκολευτούμε να βγάλουμε τα υγρά. Τα κράτη-μέλη μιλούσαν για 100 ml κατά νότα τώρα. Αλλά οτιδήποτε και να παίρνατε στο κατάστημα μέσα στα αεροδρόμια τα 125 ml. Οπότε πολύ δύσκολα ε, θα μπορούσαμε να βγάλουμε τα υγρά. Τέλο πάντων θα το συζητήσουμε το θέμα. Αλλά το βασικό που ήθελα να πω είναι αυτό που είπαμε για τα αεροπορικά ατυχήματα. Εγώ δεν το φέρω ελαφρώ το θέμα, διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίω έχουμε ασφαλεί ε, αεροπορικές μεταφορές διότι είχαμε ανεξάρτητους ανθρώπους αμερόληπτους ε, που διερεύνησαν τα ατυχήματα και δεν δεχόντουσαν πολιτικές πιέσεις για τις αποφάσεις που έπαιρναν και επικρατούσε απόλυτη διαφάνεια σε αεροπορικές μεταφορές και γι' αυτό το κοινό γνώριζε την έκβαση τη έρευνα κάθε φορά που υπήρχε ατύχημα. Οπότε, εντάξει, δεν είμαι σίγουρη ακριβώς τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά... Ε, αυτό που με θορυβεί είναι ότι αυτοί που διερευνούν έχουν συνεργαστεί με τους κατασκευαστές και με τις αεροπορικές εταιρείες κάθε φορά που σημειώθηκε ατύχημα. Τα, τους τελευταίους μήνες ε, συνέβησαν διάφορα περιστατικά και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα, αλλά θα με ενδιέφερε να γνωρίζω προς τα που κατευθύνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε ο κύριος Κούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενικέ Ρούτε, σας ευχαριστώ πολύ για τους στόχους για το επόμενο διάστημα, την επόμενη θητεία και τα κέντρα βάρους, αλλά εκεί χρειάζεται και επαρκής προϋπολογισμό. Και ε, με τρόμο διαπιστώσαμε ότι έχει περικοπεί για το 2010 ο προπολογισμό μας κατά 8,3% ιδιαίτερα για τη διευρωπαϊκά δίκτυα και προς το παρόν ε, μεγαλύτερος αντίπαλος είναι οι οικονομολόγοι. Μας λένε ότι περιορίζεται ε, η κυκλοφορία των εμπορευμάτων αφού έχουμε οικονομική κρίση σας αρκούν οι δρόμοι σας και οι χαράξεις. Τι θέλετε λεφτά εκεί. Μα δεν θα πρέπει να είναι τώρα... Ε, ένα κορβανά ο προπολογισμό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και να πηγαίνει ο καθένα και να παίρνει ό,τι χρήματα χρειάζεται για άλλου σκοπού. Θα πρέπει να είναι επαρκή η χρηματοδότηση και μέχρι τι 14 Αυγούστου νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τροπολογίε, αν δεν απατώμε. Και στη συνέχεια θα τα συζητήσουμε και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια, αλλά θέλουμε να μας υποστηρίξετε ε, ε, και όχι να γίνουν περικοπές ε, στις μεταφορές. Ευχαριστώ Δεγκράντες Πασκουάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ρέτρε που ήρθατε τόσο γρήγορα και μας είπατε τόσο ενδιαφέροντα πράγματα. Μια ολόκληρη πανοπλία θεμάτων. Πολύ σύντομα εγώ να σας πω τα εξής. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα ήταν ένα μεγάλο όνειρο, 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μετά ήταν η μεγάλη απογοήτευση, 8 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα μας ανακοινώνεται ότι αύριο θα έχουμε ανανέωση ε, των προγραμμάτων, επιβεβαίωση ή αλλαγή τους. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι στα πλαίσια της ε, ενδιάμεσης αναθεώρησης των δυσμονικών ε, προοπτικών μπορείτε να διευρύνετε αυτά τα 30 προγράμματα για τα προτεραιότητα. Στη συνέχεια, Γαλιλαίος και επιμένω, έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Αγιάλα. Και δεν είναι τυχαίο ότι συμφωνούμε. Δεν ναι, είναι δύο τα προγράμματα για το κέντρο, είναι τρία. Και εκεί πώς έχει προχωρήσει το θέμα. Και μια τελευταία ερώτηση. Τι έγινε με την εμπειρία του περίφημου σαρωτή σώματος, body scanner, που εδώ γνώρισε πολύ κακή ε, αντιμετώπιση και υποδοχή. Το έχετε επεμπολίσει αυτό ή το συνεχίζετε ως σχέδιο. Ευχαριστώ κύριε Γκράνδης Πασκουά. Κύριος Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Γενική Απευθυντά γιατί ήδη πριν από τις εκλογές είχατε αφιερώσει μία ολόκληρη ημέρα στην συζήτηση με εθνικούς συνομιλητές για το κόστος των νέων οδών κτλ. Ελπίζω ότι θα συζητηθούν περαιτέρω όλες αυτές οι προτάσεις έτσι ώστε οι οδηγοί να διευκολυνθούν και όσοι χρησιμοποιούν τα οχήματα. Πιστεύω, κύριε Διευθυντά, ότι θα πρέπει να ασχοληθείτε και με τις νέες χώρες. Με τις νέες χώρες. Υπάρχει πρόβλημα απορρόφησης κονδυλίων στις νέες χώρες όσον αφορά τις ε, υποδομές μεταφορών. Δεν θεωρείτε ότι θα έπρεπε ε, να ε, δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει εσείς, η δικιά σα Γενική Διεύθυνση, η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο να ασχολούνται με τα θέματα αυτά που είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ακόμα τρεις ομιλητές. Τι Μπιλμπάο Μπάρον Ο κύριος Κάντσι. Α, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά. Πολύ σύντομε ερωτήσεις τεχνικού χαρακτήρα. Μία ερώτηση σχετικά με την ασφάλεια που πέρα από την διάσκεψη που μας αναγγείλατε για το Σεπτέμβριο, 8 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, ε, που βεβαίως θα ασχοληθεί με όλα αυτά τα θέματα αλλά πιο επιγόντως μετά και από όλα αυτά τα ατυχήματα που έγιναν τώρα τελευταία έχει σκοπό η Επιτροπή να κάνει κάτι. Δεύτερον, στις συζητήσεις για το 2009 όσον αφορά τα πλάντεν είδα ότι ακυρώθηκαν πολλά προγράμματα, επελέγησαν πολύ λίγα είτε απερίφθησαν πολλά με επεξηγήσεις οι οποίες δεν είναι και πολύ πιστευτές. Ερώτηση. Τα προγράμματα αυτά απερίφθησαν για λόγους καθαρά δημοσιονομικούς ελήψη κονδυλίων ή υπάρχει δυνατότητα να επανεισαχθούν αργότερα ε, λόγω της συγκυρίας της κακής οικονομικής κρίσης γιατί καταλαβαίνετε ότι με 10-20% συγχρηματοδότησης ε, δημιουργείται ένας πολύ ικανοποιητικός μηχανισμός ε, για όλες τις εθνικές πραγματικότητες. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω ότι μπορούμε να επανεισάγουμε κάποια από τα ε, μία από δεχθέντα προγράμματα. Η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου είναι η εξής Ποιες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την κοινή ε, θαλάσσια πολιτική, πολιτική θαλασσίων μεταφορών. Επίσης γνωρίζομαι ότι η ανάπτυξη ιδιαίτερης ε, υποδομής ε, απαιτεί σημαντικές επενδύσεις, πράγμα δύσκολο σε αυτή τη δύσκολη οικονομική ε, συγκυρία. Κατά αυτήν την έννοια λοιπόν, ε, ποια είναι τα μέτρα τα οποία ε, θα πάρετε έτσι ώστε να διασφαλίσετε την καλή συνέχιση της ανάπτυξης των υποδομών και κάτι τελευταίο, ενδεχομένως θα ήταν καλό για όλους τους συναδέλφους και τους νέους συναδέλφους να έχουμε πληροφόρηση σχετικά με την παρούσα φάση των διαπραγματεύσεων με τις τρίτες χώρες όσον αφορά τις μεταφορές Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου, υπάρχει κάποια πληροφόρηση, αλλά εμείς θα θέλαμε πιο ενδελεχή πληροφόρηση όσον αφορά ε, αυτού του είδους ε, τις μεταφορές, κυρίως όσον αφορά τις ε, εναέριες μεταφορές. Ευχαριστώ κυρία Τικάρο. Τικάο. Τελευταία, αλλά βεβαίω όχι ελάχιστη. Η κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ρωτήσω το εξή τον κύριο Τόρ, γιατί δεν άκουσα το παραμικρό. Βρισκόμαστε σε μια οικονομική κρίση, έτσι, πανευρωπαϊκά. Ακούσαμε πολλά προγράμματα και ενδιαφέρουσε προτάσεις που θεωρώ καλό να προχωρήσουν, αλλά νομίζω ότι κανονικά θα πρέπει να κάνουμε το εξή εγχείρημα, την εξή άσκηση. Σήμερα ακούσαμε ότι ήταν πολύ μεγάλη περικοπή του προπολογισμού. Όμω πουθενά δεν βλέπω την αξιολόγηση και τον αντίκτυπο, την ανάλυση που έχουμε κάνει για το τι σημαίνουν αυτά τα προγράμματα στο πλαίσιο της σημερινής κρίσης. Μιλήσατε για τα τρία ή, e, αλλά δεν είδαμε να έχει κάνει καμιά ανάλυση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει έγκριση των προγραμμάτων. Η καινοτομία στην ευρωπαϊκή οικονομία σήμερα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει επιπλέον που εδώ στο Κοινοβούλιο έχει σταθεί ειδική επιτροπή για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Αυτή η καινοτομία λοιπόν πώς μεταφράζεται. Δεν φαίνεται σκόπιμο να έχουμε τέτοιες περικοπές τέτοιες ώρες. Στη συνέχεια. Και θα ήταν και ενδιαφέρον και αναγκαίο και ιδιαίτερα εν ώψη της κρίσης να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερος ο συντονισμός όλων των αποφάσεων που λαμβάνονται. Σήμερα στην Επιτροπή μας ακούσαμε επίσης και συζητήσαμε για την οδηγία των ευφυών λεγόμενων συστημάτων, αλλά και εκεί χρειάζεται συντονισμός ε, στο περιεχόμενο της οδηγίας με τα όσα μας είπατε εσείς σήμερα. Τρίτον, θα ήθελα να σας πω ότι στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να καταβληθεί μια προσπάθεια για να πιστούν τα κράτη για την καινοτομία αυτή ότι η μείωση του διοξιδίου του άνθρακα και το στίχημα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την οικολογία σημαίνει και καινοτομία και πρόοδο για το μέλλον. Ενώ τα κράτη μπαίνουν στον πειρασμό να κάνουν το αντίθετο. Όταν είναι οικονομική η κρίση δεν ποντάρουν προς τα εκεί τα κράτη-μέλη. Και τέλος, συμφωνώ με την κυρία Γιάλα, ανησυχούμε για την ασφάλεια στη θάλασσα. Ιδιαίτερα με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Σομαλία. Η δική μου κοινότητα, η χώρα των Βάσκων και ε, το χωριό στο οποίο ζω πλήττεται πάρα πολύ από αυτή την κατάσταση. Και θα ήθελα στους συντονιστές να ζητήσω να επιμείνουν στα προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε, κυρία Μπιλμπάου. Κύριε Ρόιτα, έχετε πάρα πολλά να απαντήσετε και δεν έχετε και πολύ χρόνο, οπότε θα, <laughs> θα συνεχίσω να κραδένω εγώ το σφυράκι γιατί σας αφορά και εσάς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ κινδυνεύω και πολύ περισσότερο γιατί είστε δίπλα μου. Ναι, χρησιμοποιώ και το αριστερό χέρι λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, ε, εν συντομία, ας αρχίσω με κάτι γενικό. Θα το πω σαφώς. Η, Επιτροπή και η, Επιτρο... η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή ε, Μεταφορών αγωνίζονται από κοινού για περισσότερα κονδύλια για τις υποδομές. Ε, πρέπει να φροντίσουμε οι επενδύσεις για τις υποδομές ε, όχι μόνο σε αυτή τη δημοσιοοικονομική περίοδο αλλά και στην επόμενη Πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να αυξηθούν τα κονδύλια γιατί πραγματικά χωλαίνει η κατάσταση ως προς επενδύσεις για τις ε, υποδομές. Ε, είχαμε την πράσινη βίβλο για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και το εγχείρημα είχε ως στόχο να προετοιμάσουμε τη μελλοντική συζήτηση για τις επενδύσεις, ε, για τις υποδομές, τις ευφυείς υποδομές, έτσι να το διευκρινίσουμε. Ε, κατά τη γνώμη μου, οι ευφυείς υποδομές ε, τι σημαίνουν. Μείωση των εκπομπών. Να μεριμνήσουμε εδώ τόσο ώστε να χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικά το σύστημα. Αυτό έχει ιδιαίτερο βάρος για το μέλλον των πολιτικών του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόεδρε, Ήδη έχω ξεφύγει σε μεγάλο βαθμό από την εντολή μου. Γιατί το λέω αυτό. Είμαι υπάλληλος, δημο... ε, ε δημόσιος υπάλληλος. Δεν είμαι ε, πολιτικός. Και ουσιαστικά λειτουργώ υπό τον έλεγχο του Αντιπροέδρου Ταγιάννη. Ε, γιατί το λέω αυτό, γιατί συζητήθηκαν πολλά θέματα μελλοντικών πολιτικών, δεν μπορώ να σας δώσω ε, απάντηση. Το κολέγιο των το σώμα επιτρόπων θα αποφασίσει. Εμείς θα δίνουμε συμβουλές ε, στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, σε όλους τους επιτρόπους. Εκείνοι όμως αποφασίζουν και εμείς στη συνέχεια υπερασπιζόμαστε τη θέση τους. Πολλές από τις ερωτήσεις λοιπόν δεν θα βρουν απάντηση από μένα σήμερα. Μπορώ να σας απαντήσω ε, για τα θέματα που σχετίζονται με τις ε, τωρινές εντολές. Εγώ πάντως μπορώ να αναφέρω αυτά που είπατε στον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Λοιπόν, για να δούμε μια σειρά από συγκεκριμένα ζητήματα που ανέφεραν ε, τα μέλη της Επιτροπής. Για, για τη μελλοντική νομοθεσία, είτε μιλάμε για μέγεθος, ε, είτε μιλάμε ε, για το κταίο, το ΤΥΒ το γερμανικό, η επόμενη επιτροπή θα αποφασίσει. Δεν είναι στο πρόγραμμα εργασίας, το τωρινό της, επιτροπής. Για το θέμα του σχεδίου δράσης και το εξάμεινο για τα αεροδρόμια και... Κύριε Ελχαντράου, δεν θα σας απαντήσω. Δεν μπορώ τώρα. Είναι σαφές ότι θα ε, συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους. Αυτό είναι σαφές. Κυρία Λίχτεμπέργε, ο Πατρίκου Ντού, από ό,τι άκουσα, θα έρθει. Που ε, ε, έκανε τον έλεγχο για τα συστήματα κράτησης ε, των παιδιών. Κατά πάσα πιθανότητα θα σας δώσω την απάντηση για τη μελέτη. Από ό,τι διάβασα, στον τύπο, έτσι, έχω, υπήρξαν κάποιες πληροφορίες, πρέπει να το εξακριβώσω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ο Πάτρικο Κοντού και υποφαινόμενος πήγαμε την περασμένη εβδομάδα στη ΣΥΠΑ και μιλάγαμε για το πιλωτικό, για, για την ε, κόπωση των πιλότων και θα το συζητήσουμε, θα συνεχίσουμε να συζητάμε το θέμα αλλά θα απασχολήσει την επόμενη Επιτροπή. Κυρία Γιάλες, ε, έχουμε την πρόταση ακόμη για τις διασυνοριακές αξιόπινες πράξεις, είναι επιτάπητος. Ας το δούμε από την οπτική γωνία του Ευρωπαίου πολίτη. Ας προσευχηθούμε να αρχίσει να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας για να ε, μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε κάτι διαφορετικό για το, για το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Υπάρχει η συμφωνία στην οποία συμμετείχα κι εγώ. Δηλαδή, θέλουμε να αρχίσει να ισχύει το κέντρο, αλλά είναι θέμα κόστους. Σαφώς ε, πάντως αυτό ήταν το αντικείμενο της συμφωνίας όπως το περιγράψετε. Ίσως δεν εξεφράστηκε σωστά για τους συντονιστές. Ε, η πρόταση που είδατε στην προηγούμενη περίοδο θα επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Σέκη θα διοριστεί ως συντονιστής. Πώς έχει συμφωνηθεί δηλαδή. Δύο συντονιστές απλά δεν θα διοριστούν γιατί ο Βαν και ο Μπαλάς δεν είναι πια διαθέσιμοι, να το πω έτσι. Για τις διαπραγματεύσεις με τις τρίτες χώρες ε, σας ενημέρω ούτως ή άλλως ε, διαρκώς και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την ενημέρωση. Δεν θα σα μιλήσω τώρα συγκεκριμένα για τι διαπραγματεύσει με το Μεξικό. Περατώθηκαν πλήρω διαπραγματεύσει με τον Καναδά. Αρχίσαμε το δεύτερο γύρο με τη ΣΥΠΑ. Και διαπραγματευόμαστε και με τις χώρες των Βαλκανίων. Θα σα ε, ενημερώνουμε διαρκώς, κυρία Τσίκα. Κυρία Μπιλμπάου, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μην αρχίσουμε τώρα γιατί θα με ακούτε για μία ώρα. Αφήστε το καλύτερα. Επί της αρχής συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει να πιέσουμε για καινοτομία, ξανά καινοτομία και κόντρα καινοτομία. Ναι, έχουν βελτιωθεί και η κατάσταση με τα οικονομικά. Εν γέννη πάντως η γάμα δέλτα τρέν έχει πολύ καλά ρεκόρ. Δηλαδή, μετατροπή της έρευνα σε συγκεκριμένα προγράμματα, ή ETMS, ε, ε, το ΣΕΖΑΡ ε, για τη διαχείριση εναέρειας κυκλοφορίας έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από όπου φαίνεται ότι αρχίσαμε με ερευνητικά προγράμματα ως γαμαδέλτα και στη συνέχεια ε, εφαρμόσαμε στην πράξη και καταλήξαμε σε προγράμματα τεχνολογικής ε, καινοτομίας. Ε, πραγματικά έχουμε πολύ ε, καλές επιδόσεις στον τομέα των μεταφορών. Κυρία Φώστερ, συμφωνώ μαζί σας για τις έρευνες για τα ατυχήματα. Πρέπει σαφώς να γίνει η διάκριση ανάμεσα στην αρχή που αδειοδοτεί για την ασφάλεια έτσι, και τις αρχές τις ερευνητικές. Ε, σωστά εντοπίσατε τις ελλείψεις ε, που υπάρχουν ε, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών, αλλά εμείς δεν συγχαίουμε αυτούς τους δύο ρόλους, είναι διακριτή. Πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη μερόληπτη αρχή διερεύνηση των ατυχημάτων. Και ίσως και χρειαζόμαστε ένα είδος δικτύου, αλλά το σκεφτόμαστε ακόμα ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Πρόεδρε, να σταματήσω εδώ. Θα σας ενημερώσω στη συνέχεια για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και το πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης ε, στους συντονιστές έτσι, που θα σας μεταφέρουν το μήνυμα. Απλά πριν ολοκληρώσω θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και τις παρεμβάσεις τους και φυσικά θα ενημερώσω τον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη για τις συζητήσεις σε uh, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Ε, επειδή έχουμε ακόμα πολλή δουλειά, ε, έχουμε την συνεδρίαση των συντονιστών, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Υπό τα διάφορα δεν έχω κάτι, απλώς να σας θυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών είναι την, ε, είναι την 3η 1η Σεπτεμβρίου, 3 το απόγευμα και στις 2 ε, Σεπτεμβρίου ελπίζουμε ότι θα έχουμε τον Γενικό Γραμματέα της ΕΑΣΑ μαζί μας. Εάν δεν θέλει κανείς να θίξει οτιδήποτε άλλο σε αυτή τη συνεδρίαση της Ολομελίας της Επιτροπής, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ και τους διερμηνείς και οι διερμηνείς ευχαριστούν τον Πρόεδρο. Ε, έκλεισε λοιπόν, τελείωσε η συνεδρίαση. Πέντε λεπτάκια για να ξεμουδιάσουμε και συνεχίζουμε. Okay,